Αγαπητοί συνάδελφοι, Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά η πολιτική ζωή τη Ευρώπη δυστυχώ δεν έχει μόνο σαν κέντρο τη την Επιτροπή Προπολογισμών. Και είχαμε συνεδριάσει, ραντεβού και με τον τύπο σε σχέση με την επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε γρήγορα γιατί είναι η εβδομάδα διακοπών για το Βέλγιο, σχολικών διακοπών εννοώ. Και επειδή είμαστε μαθητές κι εμείς, Ευρωπαϊκό Σχολείο, όλοι είμαστε Ευρωπαϊκό Σχολείο, είτε μαθητές είτε καθηγητές. Σημαντική μενει η ευρωπαϊκή επικαιρότητα, αλλά στην ημερήσια διάταξη δεν έχουμε και πολλά επίκαιρο θέματα. Έχουμε μόνο μισή μέρα. Ας τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Είδατε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε κάποια παρατήρηση για την ημερήσια διάταξη, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί. Δυστυχώς, για άγνωστους λόγους, δεν του το υφέρεις, το φταίει ποιος θέει, η κυρία Αντριάσεν δεν θα είναι παρούσα. Αναβάλλεται λοιπόν το σημείο 12. Τώρα, Ανακοινώσεις του Προέδρου. Στο Κόμπου News βλέπετε τι γλώσσες θα έχουμε σήμερα. Έχετε πρακτικά της, των εργασιών της άτυπης ομάδας για τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δύο σημεία θα επισημάνω. Το πρώτο είναι ότι έγινε το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή μιας άκρος μεγάλης σημασίας απόφαση που πήρε οικονομικής και λοιπά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Οικονομικών μετά ενέκρινε ένα μηχανισμό εφαρμογής για τον οποίο η Κομισιόν ακόμα τον επεξεργάζεται για να μετατραπεί όλο αυτό το σύνολο αυτό του πολιτικού μηχανισμού σε ένα νομικό και χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια σήμερα γιατί η Επιτροπή μας δεν είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά φυσικά θα μελετήσουμε τα διδάγματα των γεγονότων και των αποφάσεων για να δούμε τι πολιτική συνέχεια πρέπει να δώσουμε στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων μας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό οικονομικής συνεργασίας εμπεριέχει μια νέα διάσταση με βάση το άρθρο 22 της Συνθήκης Λισαβόνας, με βάση το οποίο η Κομισιόν ε, στο όνομα της Ένωσης μπορεί να δανειστεί 160 δις ευρώ για να δανείσει σε μια χώρα μέλος που θα αντιμετωπίζει εξαιρετικά προβλήματα, ανεξάρτητα της βούλησής του. Αυτό είναι μια διάσταση του προγράμματος που είναι της αρμοδιότητάς μας. Τώρα, κατά από ποιες συνθήκες, πότε με βάση ποια νομική βάση είναι νωρίς ακόμα. Γιατί όπως σας είπα η Κομισιόν τώρα που μιλάμε το επεξεργάζεται η Κομισιόν. Δεν σας προτείνω λοιπόν σήμερα συζήτηση για το θέμα. Πρέπει όμως να το συζητήσουμε. Αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο αποτελούν ένα νέο πολιτικό στοιχείο που σημαδεύει το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην οικονομική ιστορία της Ένωσης και που φυσικά για τόσες σημαντικές εργασίες όπως η προσαρμογή των δημοσιονομικών προοπτικών σε έφθετο χρόνο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Θα έχουμε ένα πρώτο ραντεβού για να το συζητήσουμε στα γρήγορα όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και με εκπροσώπους της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών ή Οικονομικών των Εθνικών Κοινοβουλίων διότι όπως ξέρετε από την 1η Ιουνίου στην 1η Ιουνίου μάλλον θα έχουμε την ετήσια συνάντηση των Επιτροπών Προϋπολογισμών της Ένωσης 1η Ιουνίου και ήδη στην εμερήσια διάταξη ως κύριο θέμα έχουμε βάλει συντονισμό δημοσιονομικών πολιτικών στην Ένωση προκειμένου να χρηματοδοτούνται καλύτερα οι κοινοί στόχοι. Αυτού που αποκαλούσαμε στρατηγική Λισαβόνας 2000-2010 και που θα είναι η στρατηγική Ευρώπη 2020 πάνω όλα πάνε καλά, θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, μετά γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Για να προετοιμάσουμε αυτή τη συνάντηση με τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, θυμόσαστε ότι επιφορτήσαμε σε ένα ειδικό γραφείο μελετών μια ειδική μελέτη συγκριτική της διάρθρωσης του προπολογισμού εθνικών και ευρωπαϊκού και το πώς σήμερα ορισμένες χώρες, γιατί η μελέτη δεν καλύπτει και τις 27, καλύπτει γύρω στις 12 χώρες. Το πώς λοιπόν αυτές οι χώρες στον προπολογισμό τους κάθε χρόνο λαμβάνουν υπόψη τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους όπως σας τα έλεγα πριν, στρατηγική σε Ευρώπη 2020. Αυτή τη μελέτη μέχρι στιγμής την έχουμε μόνο στα αγγλικά. Μεταφράζεται όμως σε όλες τις γλώσσες, σε λίγες μέρες θα την έχουμε και θα είναι έγγραφο εργασίας βασικό για τη συνάντηση αυτή. Έγκριση, σημείο 3, έγκριση των πρακτικών Τη προηγούμενη συνεδρίαση, 7 και 8 Απριλίου. Αν μέχρι το τέλο δεν έχετε σχόλια, όσοι ήθιστε, θεωρούμε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Έρχομαι στο 4. Σχέδιο έκθεσης της συζητήτρια Συντόνια για το σχέδιο προπολογισμού του 2011 Συντόνια χρειάζεται εντολή για τον τριμερή διάλογο που θα έχουμε με τα άλλα όργανα. Η συνάδελφος έχει το λόγο. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είχαν εμπλακεί στην προπαρασκευή του εγγράφου. Εργαζόμαστε υπό τεράστια πίεση χρονική για να καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε με αυτή την ταχεία μεθοδολογική προσέγγιση, ας το πω έτσι. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση για τις απουσίες μεταφράσεων και λόγω του περιορισμένου χρόνου και πάλι θα υπάρχουν σε σχέση με τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει θα υπάρξουν τα έγγραφα στη διαδικασία τη δημοσιονομική. Θέλω να επαναλάβω γιατί βρισκόμαστε υπό τέτοια πίεση χρόνου και γιατί καθυστερούν τα έγγραφα και γιατί πρέπει να εργαστούμε τόσο γοργά. Αυτό επειδή η επιθυμία μου, μια στιγμή, το όνειρό μου είναι να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο που θα εγκριθεί στην Ολομέλεια προτού γίνει η ανάγνωση από πλευρά του Συμβουλίου. Αυτό εξηγεί, επεξηγεί και ελπίζω ότι θα δικαιολογεί κιόλα ε, για αυτή την ταχύτατη διεργασία που έπρεπε να ανεχθούμε. Τώρα επί της ουσίας τι συμβαίνει. Στις 25 Μαρτίου στην ε, Ολομέλεια εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές, οι προτεραιότητες μας για το 2011 Τώρα έχουμε το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στο τραπέζι. Η δική μου έκθεση είναι σχόλιο στο σχέδιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως υποβλήθηκε σε εμά. Δεν επαναλαμβάνω λοιπόν αυτά τα οποία αναφέρθηκαν το Μάρτιο, δεν το θεωρώ αναγκαίο αυτό. Επικεντρώνομαι κυρίως σε αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Απριλίου. Τώρα, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια από τα πιο σημαντικά σημεία που όπως πιστεύω εγώ θα μπορούσαν να είναι στοιχεία κλειδιά για τον τριμερή διάλογο, για τον δημοσιονομικό τριμερή διάλογο, για τον προϋπολογισμό. Πρώτα απ' όλα η αποτίμηση, η αξιολόγηση του σχεδίου προϋπολογισμού που σαφώς δείχνει ότι τα περιθώρια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ότι ουσιαστικά δεν μας αφήνεται πλέον περιθώριο ελιγμών για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητες και στις ανάγκες μας. Αυτό δυστυχώς πρέπει και πάλι να το υπογραμμίσουμε. Πρωτού περάσω στη συζήτηση επί της ουσίας. Πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας στην παράγραφο 56 που έχει κάποια ατυχή, ας το πω έτσι, σφάλματα τυπογραφικά δακτυλογράφησης. Εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν, ε, απουσιάζουν για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση θα ήθελα να το αναφέρω να σας διαβάσω ποιο είναι το σωστό κείμενο, η σωστή διατύπωση στην πρόταση. Παράγραφος 56. Σημειώνει το 2,9% αύξησης ως ποσοστού στον διοικητικό προϋπολογισμό από πλευρά της Επιτροπής. Σημειώνει ωστόσο ότι δεν είναι όλα τα κόστη που αφορούν την διοικητική εργασία και την διπλωματική ε, υπηρεσία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη σε αυτό. Σε αντίθεση λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη σε σχέση με αυτή την παρουσίαση. Δεν θα το αναλύσω πώς συνέβη αυτό. Εγώ όμω πιστεύω ότι αυτό που έχουμε στο τραπέζι τώρα με το σχέδιο προϋπολογισμού δεν μας δίνει μια βάση για να καλυφθούν όλα τα κόστη για τη μελλοντική αυτή, τα μελλοντικά χρόνια σε σχέση με τις δαπάνες. Τώρα επί της ίδιας της ουσίας θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα πολύ γενικό σχόλιο που αφορά αυτά τα οποία <clears throat> αποκλήθηκα στην αρχή η στρατηγική για το 2020, η στρατηγική 2020 όπως την λέμε. Στην πρόταση της Επιτροπής για το Σχέδιο Προπορισμού λέγεται ότι συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική αυτή για τα προγράμματα δράσης του 2011. Εγώ ωστόσο κάποιες αμφιβολίες εκφράζω στην έκθεσή μου, γιατί μου φαίνεται ότι γίνεται λόγος για την ανα ονομασία, νέα ονομασία αυτών των προγραμμάτων, όμως υπό δημοσιονομικούς όρους δεν είναι δυνατόν για μένα να δούμε αν έχουμε περισσότερα κονδύλια για αυτές τις ναυαρχίδες, για αυτές τις, ας το πω έτσι, για αυτά τα μεγάλα προγράμματα από αυτή τη στρατηγική ή όχι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα μόνο, αλλά δεν είναι και το μόνο παράδειγμα όσον αφορά τα προγράμματα για την νεολαία, Youth Program. Τώρα έχουμε ένα νέο όνομα, Youth on the Move η νεότητα εμκινήσει, νεολαία εμκινήσει. <clears throat> Όμως ποια προγράμματα είναι εκείνα τα οποία θα ενισχυθούν και ποια βρίσκονται κάτω από αυτό τον τίτλο Youth on the Move υπό αυτή την αβαρχίδα. Λοιπόν, προφανώς αυτό πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος, να το μελετήσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Τι σημαίνει υπό όρους δημοσιονομικού, υπό τους όρους του προϋπολογισμού, η υλοποίηση δηλαδή στο μελλοντικό πρόγραμμα της, ε, στρατηγικής, ε, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020-2020. Επίσης από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα υφιστάμενα προγράμματα θα συνεισφέρουν και ποια κονδύλια, ποιοι πόροι από τα σημερινά προγράμματα θα μετατεθούν, αν θα μετατεθούν καν, και πώς θα τροφοδοτήσουν αυτή τη στρατηγική ε, για την Ευρώπη 2020. Πρέπει να παρακολουθήσουμε φοβούμε αυτό εκ του σύνεγγυς στην συνολική διαδικασία τη δημοσιονομική. Θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τοποθέτησή της για αυτό το θέμα, ή αποσαφηνήσεις. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ε, σε σχέση με την ε, νεολαία η νεότητα που είναι μια προτεραιότητα ιδιαίτερα ένθερμα την υποστηρίζω και θα πρέπει εδώ σε σχέση με το τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Αν δούμε και τους ερευνητές ε, και στο ε, πρόγραμμα για την έρευνα Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις δικές μας προσδοκίες να ενισχυθούν οι προτεραιότητες όσον αφορά την ε, νεολαία, την κινητικότητα, την, ε, ε, την παιδεία, κατάρτιση, η διαβίου εκπαίδευση. Μόνο συμβολικά έχει αυξηθεί και ούτε καν πάνω από το ποσοστό του πληθωρισμού. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα οποία αναμέναμε, δεν ήταν τα προσδοκόμενα. Όσον αφορά την κατηγορία 1β τώρα, αυτό που είναι θετικό μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια αύξηση στις πληρωμές σας είναι κάτι λοιπόν που είχαμε ζητήσει κι εμείς από την άλλη πλευρά σίγουρα και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια παράλληλη εξέλιξη σε σχέση με το πώς προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υλοποίηση αυτής της συνιστώσας. Το πολιτικό μας αίτημα για την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και ελπίζω ότι θα ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό και αυτό με κάνει να καλωσορίσω αυτή την αύξηση στις πιστώσεις πληρωμών. Για την κατηγορία 2 τώρα είναι σημαντικό να πούμε να αναφέρουμε ότι υπό την συνθήκη της Λισαβόνας και τα δύο σκέλη της δημοσιονομικής αρχής θα έχουν ίση, ίσο μερίδιο, ίδιο μερίδιο αρμοδιοτήτων και εξουσιών, αλλά και περιορισμούς εξίσου. Και θα ήθελα εδώ για την ε, ε, από συνδεδεμένη υποστήριξη και να υπενθυμίσω ότι για την Ολομέλεια δεν ήταν δικό μου αίτημα, αλλά από κάποιους ευρωβουλευτές το Μάρτιο είχε ζητηθεί να συζητηθούν προγράμματα που συνδέονται με το γάλα στα σχολεία και τα ε, ε, οποροκυπευτικά στα σχολεία και σημαντική αύξηση αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημειώνω αυτό και είναι μια καλοδεχούμενη εξέλιξη. Μετά υπάρχει και μία αύξηση όσον αφορά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Είναι μία ευπρόσδεκτη εξέλιξη και αυτή. Επίσης ε, έριξα μια ματιά στο τι γίνεται με το Frontex, μια επικαιροποίηση αυτών που τεκταίνονται και αυτά που είδαμε όσον αφορά τις αδυναμίες, όσον αφορά την εκτέλεση των μέτρων από πλευράς ε, ε, Frontex. Τώρα σε σχέση με την κατηγορία 4, εδώ πρέπει και έπρεπε να εκφράσω την ανησυχία μου. Και αυτό για την μείωση των κονδυλίων για την Παλαιστίνη. Είναι κάτι, πιστεύω αυτό, που πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, πιο προσεκτικά. Και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα αυτή η μείωση. Και σημείωσα για την στρατηγική, για την ε, Βαλτική, ε, είναι και αυτό σημαντικό θέμα για την ε, στρατηγική μας. Για την κατηγορία 5 τώρα. Αυτό που είδα στην κατηγορία 5 το ερμηνεύω ως μια κίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφήσει ένα περιθώριο που θα έδινε δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όσον αφορά την ευρωπαϊκή εξωτερική ε, υπηρεσία. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα να απαντηθούν εδώ το περιθώριο είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να είναι ένα αντικείμενο συζήτησης για τον τριμερή διάλογο. Επίσης με ανησυχεί κάπως το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβλεψε κανένα κονδύλιο για τα πιλωτικά προγράμματα για την προπαρασκευαστική δράση. Είναι προμεμόρια, προμεμόρια PM, προσυπόμνηση και αυτό είναι θέμα για μας το φθινόπωρο να αξιολογήσουμε και να δούμε αν θα δοθεί συνέχεια σε αυτές τις προπαρασκευαστικές δράσεις ή πιλωτικά προγράμματα. Αφήνει αυτό ένα περιθώριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουμε, να δούμε αν θέλουμε να συνεχιστούν αυτές οι δράσεις ή όχι και να τοποθετηθούμε αντίστοιχα. Τώρα, σε αντίθεση με την πρακτική από προηγούμενα χρόνια, δεν επέλεξα κάποια από τα ε, θα έλεγα προτιμόμενα θέματα για τον κατάλογο, για τον τριμερή διάλογο, θα έπρεπε να έχουμε εμεί την ελευθερία τελικά να είμαστε σε θέση κατά τον τριμερή διάλογο να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε ένα από τα σημεία που προκαλούν ανησυχίες και που έχουμε εντοπίσει, έχουμε ταυτοποιήσει. Σύμφωνα με μένα κάθε σημείο του σχεδίου εντολής θα μπορούσε να είναι, δεν πρέπει υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα σημείο που μπορεί να τεθεί υποσυζήτηση στον τριμερή διάλογο. Εδώ θέτω μια άνω σταματώ και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Συντόνια. Σημειώσουμε το ότι πρέπει να, προσθέσουμε το σημειώνεται. Ο φίλος μας ο Τζέιμς Έλλης κάποια στιγμή παλιότερα με βάση έναν Άγγλο χιουμορίστα. Όταν μια lady λέει not, not, όχι, not, σημαίνει ίσως. Όταν λέει ίσως σημαίνει ναι. Αν πει ναι δεν είναι lady. Άρα σημειώνουμε εδώ not, όχι. Όταν η συντονία λοιπόν δεν λέει τίποτα, αυτό σημαίνει not, not. Είναι καλό αυτό για έναν εισηγητή του προπολογισμού να λέει όχι να μπορεί να λέει όχι. Έλλης. Το αντίθετο είναι ο διπλωμάτης είναι ακριβώς το αντίθετο. Το διπλωμάτης ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή όταν ο διπλωμάτης λέει ναι σημαίνει ίσως, όταν λέει ίσως σημαίνει όχι και αν είναι όχι δεν είναι διπλωμάτης. Συμφωνούμε. Πάντως οι του προπολογισμού πρέπει να λένε όχι πάντα. Πάντα αλλά υπάρχει το ανόητο όχι και το έξυπνο όχι. Και προσπαθούμε να λέμε όχι έξυπνα. Σας προτείνω να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν και μετά ο Γενικός Διευθυντής του Προϋπολογισμού που μας ε, περιπείται την τιμή να συμμετέχει στην συνεδρίασή μας θα απαντήσει και αυτός στα ερωτήματα της εισηγήτρες και των συναδέλφων. Η κυρία Μπαλτσάνη. Ευχαριστώ. Η Συντόνια κάνει μια δουλειά πάρα πολύ ακριβή και χρήσιμο είναι να την υποστηρίξουμε σε αυτό το λεπτό και δύσκολο πέρασμα που ζούμε. Ωστόσο, υπάρχουν προσαρμογές που θεωρώ χρήσιμες σε αυτή τη φάση στο έγγραφο εντοκής. Πρώτον, στις γενικές παρατηρήσεις θα πρέπει να ξανατονίσουμε την ανάγκη μιας βαθιάς αναθεώρησης των οροφών των δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό που έγινε αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες θα έλεγα, καθιστά σκόπιμο να υπογραμμίσουμε τη σημασία μιας ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση και στις νέες ανάγκες. Την ανάγκη συνεπώς μια, πιο μεγάλου προπολογισμού της Ένωσης με μεγαλύτερη ευελιξία. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και στο κείμενο αυτό. Μεταξύ των προτεραιοτήτων, πέρα από το, θέμα νεότητα και σημασία της, που το τονίσαμε ειδικά όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες, καλό θα είναι στις γενικές παρατηρήσεις, general remarks, να επισημάνουμε τη στρατηγική 2020 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να είναι σκληρή, να επιβάλλει κυρώσεις κατά κάποιο τρόπο σε χώρες που δεν θα υιοθετήσουν μέτρα προκειμένου να γίνονται πράγματα σε αντίθεση με αυτό που δεν έγινε με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Επειδή όμως μιλάμε για εντολή και για μια νέα διαδικασία προϋπολογισμού, το Κοινοβούλιο πρέπει να τονίσει την αποφασιστικότητά του να αποφευθούν μαθηματικές λύσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να ορίσουμε πολιτικές προτεραιότητες, χρήσιμες, διαφανείς, ορατές. Δεν μπορεί να δοθεί μαθηματική απάντηση που να μην λαμβάνει υπόψη αυτή την προσπάθεια του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έργα σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θυμάστε όταν ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι παρουσίασε το σχέδιο προπολογισμού για την Κομισιόν μα έδωσε και μια αφίσα που με χαροποίησε ήδη από τις 28 Απριλίου γιατί ήταν αφίσα από τις ε, προεκλογική αφίσα των Πρασίνων με το όνομα Green New Deal. Θυμάστε τέσσερις στήλε, μία ήταν πράσινη. Αυτό το οποίο είχαμε πει δηλαδή πως ε, πρέπει να αλλάξουν οι προϋπολογισμοί με τους ε, διάφορους ε, τομείς, να αλλάξει δηλαδή η πολιτική της παιδείας, της έρευνας, της γεωργίας, της διαρθρωτικής και κάποια άλλη τομείς και βεβαίως πάνω απ' όλα η αλλαγή του κλίματος. Και είναι ενδιαφέρον τώρα πως ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι για τον προπολογισμό του, του 2010 11, ε, επέλεξε την πράσινη πρόταση. Και λέει βεβαίως πως ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι πράσινος. Αλλά πού στηρίζεται αυτό. Ας δούμε τα νούμερα και την ουσία. Το τι δηλαδή θα είναι πράσινο με την έννοια της οικολογικής και αηφόρου αλλαγής. Όσον αφορά την γεωργία, οι κύριες ε, πληρωμές πάνε στις, ε, στη στραματική ενίσχυση. Οπότε δεν το βλέπουμε αυτό κάπου. Είχαμε κάνει όμως το check-up και έχουμε και αυτά τα οποία μας προτείνουν οι μελέτες του ΩΣΑ, πως δεν είναι αρκετά η η πολιτική γεωργίας και πως θα πρέπει παραδείγματος χάρη να συνδεθούν οι πληρωμές με παραγωγή οικολογικής ενέργειας με τα διαρθρωτικά ταμεία. Το ίδιο πρόβλημα. Εάν δούμε και αν παίρνουμε όντω στα σοβαρά την πολιτική προστασία του κλίματο, θα πρέπει να ανακαινήσουμε ενεργητικά τα κτίρια μα, έτσι ώστε να μπορούν να εκπέμπουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε ούτω ή άλλω δηλαδή, αν παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μα, όχι μόνο για τον προπολογισμό του 2011. Διαπιστώνουμε όμω εδώ πέρα πω τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορός, κατά βάση πάλι μιλάμε για δρόμους, αεροδρόμια και άλλα τέτοια συγκοινωνιακά έργα. Έχουμε μία αύξηση κατά 16,8% και στη διαβίου κατάρτιση όπου πάντα εξακολουθεί να μας λέει η δεύτερη επιτροπή Μπαρός όπως πρέπει να κάνει ακριβώς εκεί πέρα περισσότερα πράγματα να εκπαιδεύσει τους νέους έχουμε μια αύξηση μόνο 2,6% οπότε διαπιστώνω ότι σε σχέση με την παραδοσιακή πολιτική γεωργίας και συγκοινωνιών πως εξακολουθεί να υπάρχει μια ανισορροπία. Το ίδιο διαπιστώνω και στο θέμα της περαιτέρω μείωσης ε, των ε, εξαγωγικών επιστροφών που θα έπρεπε να εξαφανιστούν πιο γρήγορα γιατί γνωρίζουμε πως με αυτή την επιδότηση των γεωργικών μας προϊόντων ε, εξολοθρεύουμε τις αγορές της Αφρικής. Επίσης να αναφέρω την αηφορία της πολιτικής αλληλείας. Και εκεί πέρα έχουμε έγγραφο της Κομισιόν που διαπιστώνει ρητός πως έχει αποτύχει η πολιτική της αλληλείας γιατί δεν είναι αηφόρος. Και αυτό θα ήθελαμε να το δούμε στον προπολογισμό του 2011, γιατί έχουμε λάθος εδώ πέρα. Αν δεν, αλλάξουμε, αν δεν αρχίσουμε να αλλάζουμε την πολιτική, χάνουμε τον χρόνο για τα απαραίτητα βήματα αυτά. Γι' αυτό το βρίσκω λυπηρό το ότι δεν γίνονται περισσότερα και θα έπρεπε να, είμαστε, να δώσουμε εντολή στην διαπραγμάτευση για τον τριμερή διάλογο, να δοθεί περισσότερο βάρος στην αηφορία και στην οικονομική ανακαμψή. Να φέρω κάποια ακόμα ερωτήματα που ε, αφορούν έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Στο μεγάλο τίτλο νεολαία εγκινήσει, κατά την άποψή μου δεν τονίζεται αρκετά πως θα πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους νέους και όχι μόνο σε αυτούς με την ανώτατη εκπαίδευση. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό όσον αφορά και την πολιτική αποδοχή του στην Ευρώπη. Όλοι δηλαδή θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία για περισσότερες ανταλλαγές και κινητικότητα. Ίσως λοιπόν η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει ένα ερώτημα και στην ε, τωρινή πρόταση Αναφέρθηκε ήδη πως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα για τα σχολεία. Όμως στην ε, κάτω Σαξονία και στην Βρέμη το πρόγραμμα αυτό για τα φρούτα στα σχολεία ε, βρήκε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση, πάρα πολύ κακά δημοσιεύματα και νομίζω υπονόμευσε τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα μπορούσε η Κομισιόν γραπτός ίσως να μα πει ποιο είναι το πρόβλημα που θεωρεί εκείνη ότι υπάρχει στην εφαρμογή για να μην υπάρχει πλέον αυτή η αντίδραση και η οργή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σαλβατόρ Γκαρίγα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπατε για το πώς λέει κανείς έξυπνα όχι ή με έτσι πιο χοντροειδή τρόπο. Δεν ξέρω εάν το ναι θα πρέπει να είναι, το όχι με συγχωρείτε θα πρέπει να είναι σε μια εντολή τριμερούς ε, διαλόγου. Τώρα ελπίζω λοιπόν να το όχι που θα πούμε εμείς να είναι υπό όρους. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στον ε, τριμερή αυτό διάλογο έτσι ώστε το όχι να καταστεί ναι και να μην έχουμε το συντομότερο τριμερή διάλογο στην ιστορία. Γιατί η συμφωνία για τους ε, τροποποιητικούς ε, αυτούς προϋπολογισμούς είναι απαραίτητη. Πρέπει επίσης να έχουμε ένα σχέδιο για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που βεβαίως θα διευκολύνει την εισηγήτρια και πιο εύκολη το έργο της συνδιαλλαγής για αυτή την Επιτροπή Προϋπολογισμού, για αυτόν τον τριμερή διάλογο. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τώρα το μπαλάκι είναι στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι όσο θα προσεγγίζει αυτός ο τριμερής διάλογος θα έχουμε θετικές ειδήσει ε, ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα στην, διαπραγματευσή. Υπό το πρίσμα της ε, έκθεσης της Ιδόνια εν πάση περιπτώσει είναι συμπέρασμα, είναι αυτό, αυτά που έχουμε εγκρίνει στις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό. Και τώρα με την εντολή να μεταφραστούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές σε μια σαφή στρατηγική διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο σε αυτόν τον πρώτο τριμερή διάλογο και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι την υποστηρίζουν στην έκθεση που μας έχει παρουσιάσει και μπορεί και ίσως ακόμα να κατατεθεί κάποια τροπολογία για να ισχυθεί το ένα ή άλλο σημείο. Θα ήθελα κάπως να τονίσω περισσότερο το θέμα των flagships, των ναυαρχίδων, των σημαντικότερων εγχειρημάτων που θεωρώ ότι αποτελούν το πιο καινοτόμο τμήμα της παρουσίασης ε, που έγινε από πλευράς ε, του κυρίου Λεβαντόσκη στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην ε, αναφορά που έκανε και η ίδια η Συνδόνια επ' αυτού. Εδώ έχουμε μια πρώτη ποσοστοποίηση από πλευράς προϋπολογισμού του τι σημαίνει η στρατηγική 2020 <clears throat> και μέσα σε αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να αποσαφινιστεί ότι αυτές οι πολιτικές, αυτά τα θέματα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ως θεμελιώδες τμήμα αυτής της στρατηγικής. Με άλλα λόγια, μέσω του προϋπολογισμού του 2011 θα έχουμε μια σαφέστατη ένδειξη για το ποια θα είναι η στρατηγική του 2020 και οι δεσμεύσεις από πλευράς προϋπολογισμού των κονδυλίων δηλαδή που θα πρέπει να εξεταστούν όπως ανέφερε η κυρία Συντόνια σήμερα είναι ε, ουδέτερες δημοσιονομικά πολιτικές σε σχέση με το, τη διαμόρφωση του προπολογισμού 2011 δεν αποτελούν σήμερα μια επιλογή όσον αφορά ξεχωριστή δυνατότητα. Και αν αληθεύει ότι μέσα σε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 θα έχουμε μια ένδειξη για αυτές τις ναυαρχίδες flagships, τώρα πλέον είναι σαφές ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει πλέον την πολιτική επιλογή και εναλλακτική λύση να αλλάξει, να τροποποιήσει την ίδια τη σύνθεση θα έλεγα των τμήματων της στρατηγικής 2020 και από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την επισήμανση των θεμελιωδών στοιχείων αυτής της στρατηγικής που εξετάζονται μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού. Είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, σε σχέση με το εγχείρημα του προϋπολογισμού του 2011 και ακόμα πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, ο, ρόλ, ρόλος από πλευρά του εισηγητή επί του προπολογισμού και τέλος πάντων έχουμε αρκετές προκλήσεις ε, και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στους επόμενους μήνες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική 2020 που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Επιτροπής Προϋπολογισμού το κάνει πιο θελκτικό ακόμα αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είχα την ε, δυνατότητα να εργαστώ λίγο καιρό επ' αυτών των γραμμών το, του προπολογισμού. Και υπάρχει εδώ πέρα μια διαφορά μεταξύ της δικής μου ανάλυσης και αυτών που αναφέρει η Συγγετρία και τα στοιχεία 2007, 2008, 2009. Πρώτα απ' όλα, αν μιλήσουμε για τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων. Έχουμε πράγματι μία μικρή αύξηση 0,7%, αλλά αν δούμε το 2009-2010 είχαμε μείον 0,8% και δεν είναι 6% το 8-9% και ούτε 9% το 7-8 συνολικά. Οπότε φαίνεται πως δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε περισσότερες ε, πιστώσεις ε, τόσο γρήγορα όσο είχαμε κάνει στην αρχή των δημοσιονομικών προοπτικών. Εάν τα δούμε τώρα αναγραμμή, και ξέρω αυτές ε, οι οποίες αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα και αυτές που είναι στο μείον, θα ήθελα να σχολιώσω πως ε, έχουμε 19% αύξηση στις, ε, στα οικονομικά και νομισματικά ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνο στο 2%. Στη δε επιχειρηματικότητα έχουμε το αντίθετο, έχουμε μείον 88% και Εάν δούμε τα 600, 655 εκατομμύρια και αν δούμε ακριβώς ποιο ήταν το μεγαλύτερο ποσό, ήταν το Γαλιλαίο και το Έγνος στην δορυφορική ε, ναυτιλία. Μιλάμε για μείον 700 εκατομμύρια, οπότε δεν πληρώνουμε για αυτά πλέον. Επίσης αυτό το οποίο είπε η συγγήτρια είναι σωστό. Συμβολικά π.χ. το Εράσμους για τους ε, νέους επιχειρηματίες είναι μείον 3 εκατομμύρια, αλλά είναι μείον 60%. Ε, μιλάω πάντα εδώ πέρα για τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων. Επίσης μετά στη Γεωργία υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια να ανακτήσουμε αυτές τις ε, υποχρεώσεις. Καθώς 9-10 είχαμε μείον 3,3%. 2 δισεκατομμύρια, κυρίως στην αγροτική ανάπτυξη. και προσπαθούμε επίσης να ανακτήσουμε 0,1% οπότε κατ' ουσίαν μένουμε στο 0. Δεν είναι εύκολο και για όσους θεωρούν πως η ενέργεια είναι το, το μέλλον, είναι σαφές εδώ πέρα στον προϋπολογισμό. Τα ενεργειακά έργα είναι ενός και δύο ετών, οπότε υποχρεώσεις για νέα δίκτυα και αποθήκευση άνθρακα κτλ. Αυτό είναι φέτος και τέλος. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τις υποχρεώσεις. Το σχέδιο ανάκαμψης είχε συνδεθεί με την ενέργεια και δεν συνεχίζεται το 2012, 2013 και 2014 σύμφωνα με αυτόν τον προπολογισμό. Επίσης ε, και ψαράς αν ήμουν δεν θα ήμουν πολύ ικανοποιημένο γιατί και εδώ πέρα έχουμε κάπως μικρότερες υποχρεώσεις κατά 0,5% και στην, ε, στις δε διεθνεί ε, αλευτικέ συμφωνίε έχουμε μείον 6%, ε, 54 εκατομμύρια. Εσωτερική αγορά επίσης, 25% αύξηση, κάτι το οποίο είναι θετικό γιατί έχουμε μέτρα τα οποία αυξάνουν, ε, βελτιώνουν την αγορά. Στην περιφερειακή πολιτική είναι σαφή τα πράγματα, έχουμε 4% αύξηση, μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο γιατί έχουμε τη συνοχή τώρα, αλλά βλέπουμε και 13% αύξηση των ε, υποχρεώσεων στον ε, τομέα της εκπαίδευσης. Σωστό. Τώρα για την υγεία και προστασία των καταναλωτή είμαστε στο μείον και είμαστε στο μείον για δύο χρόνια. Στο 9-10 ήμασταν 2% ε, μείον και το 10-11 είμαστε 3,3% μείον. Δεν είναι μεγάλα τα νούμερα. Επίσης προγράμματα καταπολέμησης ζωονόσων δεν είναι μεγάλα τα νούμερα, αλλά έχουμε αναλογικά μειώσει. Επίσης για την ασφάλεια, εγώ ήμουν και υπουργό εσωτερικών, ε, ένα είναι σαφές, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις ε, υποχρεώσεις που έχουμε για το σύστημα πληροφοριών Schengen 2 και είναι κρίμα γιατί έχουμε 14% λιγότερα κονδύλια, αλλά ανταυτού δεσμευόμαστε να δώσουμε περισσότερα, 30% περισσότερα στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, 22% περισσότερα σύνορα και πολύ περισσότερα για ένταξη υπηκών τρίτων χωρών, 21 εκατομμύρια παραπάνω. Τώρα, οι εξωτερικές σχέσεις, σύμφωνα με τον προπολογισμό, οπωσδήποτε θα συζητηθούν στην Επιτροπή Εξωτερικών, γιατί βλέπουμε πως για την Παλαιστίνη έχουμε 30% λιγότερες πιστώσεις υποχρεώσεων. Για τις ανατολικές ε, χώρες έχουμε αύξηση 20% και για τη συνεργασία με το Αφγανιστάν, με την Ασία και το Αφγανιστάν έχουμε συν 25%. Ένα είναι σαφές ε, ε, αναπτυξιακή συνεργασία με χώρες Αφρικής, Καραβικής, Ειρηνικού. Έχουμε μείον 5% αλλά καλύτερα είναι από πέρσι που είχαμε μείον 28%. Και τέλος πρέπει να πω πως ε, η ενέργεια, το είπα ήδη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί το 2010 αλλάζουν οι γραμμές του υπερπολογισμού, σπάει η ενέργεια και δεν πάει μαζί με τις μεταφορές και οι μεταφορές πάνε μαζί με την κινητικότητα. Αν δούμε λοιπόν μεταφορές και κινητικότητα έχουμε αύξηση κατά 10% και η έρευνα για την ενέργεια, δόξα του Θεώ, έχουμε κατά 27% αύξηση των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων. Αλλά τα μεγάλα έργα τελείωσαν. Και τέλος πρέπει να πω πως ε, όπως έχει γράψει η συγκήτρια, για τις ε, πλήρωμες είναι μεγάλη η διαφορά, γιατί όπως λέει και η συγκήτρια, η διαφορά μεταξύ υποχρέωσεων και πληρωμών θα γίνει πολύ μικρότερη. Έχω και άλλα σχόλια για τις ε, πληρωμές. Υπάρχουν κάποιες πληρωμές οι οποίες ε, μειώνονται σοβαρά και τέλος πρέπει να συμφωνήσω με την εισηγήτρια «90% προπαρασκευαστικών έργων είτε έχουν ε, τελειώσει είτε είναι στο απόθεμα». Έχουν τελειώσει λοιπόν αυτά τα έργα ή δεν υπάρχει τα πιλωτικά έργα έχουν τελειώσει, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν κονδύλια να ολοκληρωθούν. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί εκεί πέρα πραγματικά έχουν λεξιτοποιηθεί τα κονδύλια. Σε ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφοι. Πολύ σημαντικά τα νούμερα που ανάφερε. Η συνάδελφο Γκρέσλε. Ε, ευχαριστώ. Αν δούμε το πώς ε, πώς ανισχούν οι πολίτες μας, οι ψηφοφόροι μας για το ευρώ. Θεωρώ πως ε, θα πρέπει λίγο να ασχοληθούμε με αυτή την ανησυχία και να δούμε τελικά ποιος τηρεί και ποιος δεν τηρεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μιλάω εδώ πέρα βεβαίως για τα κριτήρια σταθερότητας που αφορούν ε, όλες τις ε, χώρες και αν θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποια πράγματα περαιτέρω για την ε, αηφορία στην ε, εντολή, νομίζω θα έπρεπε να, να ασχοληθούμε. όπως σας είπα, ποιο τηρεί και ποιο δεν τηρεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το ισχυρό μας σημείο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν νομίζω μηχανισμοί που επιτρέπουν να το εξετάσουμε αυτό τακτικά και να αντιδράσουμε. Και εγώ πραγματικά κατηγορώ και τον εαυτό μου για το ότι δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Πρώτη παράκληση αυτή, θα ήθελα λοιπόν να το, το σκεφτείτε. Εάν δεν αντιδράσουμε τώρα εδώ μέσα, τότε τελικά θα έχουμε και σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας ε, με τους ψηφοφόρους μας. Θα μας ρωτήσουν τι κάνατε. Δεύτερον, εξωτερική πολιτική. Βλέπουμε εδώ πέρα πως το μέσο σταθεροποίησης ε, το οποίο θέλει να το ενσωματώσει η εξωτερική υπηρεσία και έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, 32%. Αναρωτιέμαι μήπως ε, κάνουμε καλά ε, τα προγράμματα αυτά τα οποία υπό όρους πάνε στην ε, εξωτερική πολιτική, να δούμε πώς θα διαχειριστούν από ποιον και πώς ή αν θα έπρεπε έτσι να το αφήσουμε έτσι να περάσει τόσο εύκολα. Αυτό το ICI είναι 30% συν 32% στο μέσο σταθερότητας ή το, το πρόγραμμα πυρηνική ασφάλεια που επίσης είναι στον κατάλογο αυτό αν θέλετε των επιθυμητών. Να δούμε δηλαδή τι είναι έξυπνο για μας να κάνουμε και να υπάρχει και μία... Να βλέπουμε και κάπως το μέλλον στον προϋπολογισμό, να δούμε πώς το προγραμματίζουμε. Επίσης, το τι προγραμματίζεται να γίνει με αυτά τα, τα κονδύλια, τι δικαιολογεί αυτή τη μεγάλη αύξηση. Αυτό ισχύει π.χ. και για το συν 16% στον προπολογισμό εξωτερικών. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει και εδώ πέρα κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζω. Ευχαριστώ. Oui, le respect Ευχαριστούμε, Ο σεβασμός των κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να μας απασχολούν. Η απάντηση στο ερώτημα της ΣΥΝΚΙ είναι απλή. Καμιά από τις 20. 27 χώρες δεν το σέβεται αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Έκτακτη κατάσταση. Πάντως το θέμα αυτό, αν θέλουμε να συμβάλλουμε, να δώσουμε ένα input κι εμείς, θα πρέπει να συντονιστούμε με την Οικονομική Επιτροπή που παρακολουθεί το θέμα αυτό. Τρεις συνάδελφοι ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Φέρουν πρώτος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω, όπως και πολλοί άλλοι, ότι πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση αυτή. Βρισκόμαστε πολύ κοντά, θα έλεγα, σε μια ευρεία συνένεση απόψεων για τις πολιτικές και προτεραιότητες μας. Νομίζω η Συντόνια έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, θα ήθελα κάποια λίγα σχόλια να κάνω. Ιδιαίτερα όσον αφορά γενικό σχολιασμό αυτό του πρώτου τη έκθεση. Θέλω να υπογραμμίσω αυτά που αναφέρθηκαν πιο πριν. Τρει παραγράφου έχουμε για πολιτικέ προτεραιότητε εδώ. Την παράγραφο 7 που αναφέρεται στι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι παραγράφου 8 και 9 προτεραιότητε ε, του Ευρωκοινοβουλίου και οι δύο για την νεολαία, για την νεότητα και ναι, νομίζω πολύ καλά αυτές οι προτεραιότητες. Όμως η κυριότερη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Για την στατική για το 2020 ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης και αηφορία. Αυτό θα ζητούσε, θα απαιτούσε να έχουμε κάποια εδάφια που να αναφέρουν ότι αυτή είναι η κύρια προτεραιότητά μας και πρέπει να το συμπεριλάβουμε αυτό πιστεύω. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθούμε και όλοι το ξέρουμε ότι το κύριο πρόβλημα εφέτος θα είναι τα οικονομικά προβλήματα των κρατών μελών που οφείλονται στην κρίση, η διστακτική θέση τους ε, όσον αφορά την αύξηση τη συνεισφορά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα και πρέπει εδώ ευθύ εξ αρχή να το αναφέρουμε. Ιδιαίτερα υπογραμμίζοντα αυτά που εσύ, Πρόεδρε, έκανε πολλέ φορέ, την ανάγκη δηλαδή να αναφέρουμε, να τονίσουμε, να υπάρξει πρόσθετη αξία <clears throat> στον προπολογισμό όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, αλλά και ο συμπληρωματικό χαρακτήρα μεταξύ εθνικών προπολογισμών και ευρωπαϊκού προπολογισμού. Αυτό πρέπει να δώσουμε ω κίνητρο στα κράτη-μέλη, ακόμα και όντα σε μια χρηματοοικονομική κρίση, τα κράτη-μέλη να μπορούν να δουν αυτή την προοπτική τη ε, σωστή χρήση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Να το τονίσουμε αυτό στις, ε, στην αρχική παράγραφο για να αποφύγουμε επικρίσει ε, όταν θα έρθει η ώρα να απαιτηθούν περισσότερα κονδύλια για ευρωπαϊκέ πολιτικέ αρχή λοιπόν να ενισχύσουμε θα έλεγα αυτή την άποψη από πλευράς Ευρωβουλής θέτοντας αυτές τις πολιτικές προτεραιότητες ως Ευρωκοινοβούλιο. Και έχω και μια ερώτηση προς τη Συντόνια. Μεθοδολογική περισσότερο αυτή η ερώτηση. Είναι μια εξαιρετική έκθεση αυτή η Συντόνια. Σίγουρα. Το πιστεύω αυτό. Είναι πολύ καλή η έκθεσή σου. Όμως πιστεύω ότι μια και εμπεριέχει 73 παραγράφους και θα καταλήξουμε και σε περισσότερες στην τελική διατύπωση, δεν μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις παραγράφους στην ημερήσια διάταξη για τον τριμερή διάλογο. Κάποτε σε κάποια φάση χρειάζεται μια σε μεγαλύτερο βάθος συζήτηση για το ποιε ποιε είναι οι πραγματικέ μας προτεραιότητες Δηλαδή, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη. Ποιε είναι οι προϋποθέσεις, οι όροι μας και ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ ε, για αυτή την πολιτική ε, προσέγγιση της διαπραγμάτευσης Με ποιο πνεύμα πρέπει να γίνει. Και εν μέρη θα πρέπει αυτό, αυτή η δουλειά να γίνει και κλεισμένων των θυρών για να μπορέσουμε να βρούμε την σωστή κατεύθυνση για τις προτεραιότητες μας επίσης πιστεύω, και αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου, ότι πρέπει να προβληματιστούμε κάπω να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε τις άλλες εξειδικευμένες συγκεκριμένες συνεμπλεκόμενες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ε, <clears throat> και όταν έχουμε ως ήθιστε τις γνωμοδοτήσεις από πλευρά τους ε, και όταν θεωρείτε ότι καλύπτονται μέσω κάποιων τροπολογιών αυτά τα θέματα, όμως αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Είμαστε σε πρώτη φορά σε αυτή τη νέα διεργασία, έχουμε πάντα τονίσει ιδιαίτερα ότι χρειαζόμαστε πραγματική συνεργασία, αυθεντική συνεργασία με τις εξειδικευμένες αυτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και γνωρίζω ότι λόγω, λόγω περιορισμού ε, χρονικού δεν, είχα, δεν είχαν τοποθετηθεί όπως θα, όπως θα έπρεπε σε αυτή την έκθεση, αλλά να ακούσουμε τις απόψεις τους, είτε πρόκειται είτε αν έχουν συνυπογράψει ε, τροπολογίες ε, μέσω των ε, εισηγητών θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη δική μας τοποθέτηση τι δικέ του απόψει για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω για αυτή τη διαδικασία αν έχει προβληματιστεί σχετικά η συντόνια γιατί είναι και αυτό κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Ευχαριστώ κύριος Μπόκρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τον Γέρεν και με κάποιους άλλους που τόνισαν την ε, σημασία του να είναι ξεκάθαρες οι προτεραιότητές μας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω μία από τις σημαντικότερες, αν όχι την σημαντικότερη προτεραιότητα φέτος, την καταπολέμηση της κρίσης δηλαδή. Έχοντας διαβάσει το έγγραφο της Κομισιόν, έχει χάσει τον στόχο καθώς μιλάει σαν να έχουμε, περάσει, να έχουμε ξεπεράσει ήδη την κρίση. Κι όμως είμαστε ακόμα εν μέσω της κρίσης η οποία μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερη. Τώρα, όταν υπάρχει κρίση, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να το αντανακλά αυτό. Μπορούμε ακόμα και να τον ονομάσουμε προϋπολογισμό κρίσης. εθνικοί προϋπολογισμοί ξαναγράφονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να καταπολεμήσουν ακριβώς την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε πως ε, μάλλον το σημαντικότερο μέσο, μέτρο θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξαναβρούν δουλειά. Και πρέπει εδώ να είμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι ε, από όσο πρότεινε η κυρία Γεντρέζευσκα. Τύχει αν δούμε αυτή την πρωτοβουλία νεολαία εν κινήσει, που είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020, αυτή τη στιγμή ε, είναι μόνο ένα σύνθημα. Σε σύγκριση με το τι έχουμε στα υπάρχοντα προγράμματα. Οπότε δεν θα δώσω πολύ ε, βάρος σε αυτό αλλά υπάρχει ένα άλλο που λέγεται νέε δεξιότητε και δουλειέ θέσει εργασία. Αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Με ή χωρίς να ενισχύσουμε περαιτέρω τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια είναι σε κακή κατάσταση και για την βελτίωσή τους το θέμα είναι όχι πόσα περισσότερα χρήματα θα ξοδέψουμε, αλλά πώς θα αλλάξουν οι δομές διοίκηση εσωτερικέ και εξωτερικές. Αλλά όταν μιλάμε για νέε δεξιότητες και δουλειέ. αυτό πραγματικά είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι στο οποίο θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια, αρκεί βεβαίω να υπάρχουν μηχανισμοί για να διασφαλίσουμε πως ε, τα λεφτά που θα ξοδέψουμε εκεί πραγματικά θα ενισχύσουν τις δεξιότητες όσων χρειάζονται να ξαναπάνε να δουλέψουν. Ειδικά να σκεφτούμε το μέλλον της ε, Ευρώπης, ε, τότε προφανώς η ανεργία των νέων είναι θεμελιώδης αδυναμία αυτή τη στιγμή. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι πολύ μικρός, γνωρίζω πως δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που μπορούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί αλλά τουλάχιστον η δομή και οι προτεραιότητες του δικού μας προϋπολογισμού μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα στους εθνικούς προϋπολογισμούς, το πώς βλέπουμε εμείς αυτές τις προτεραιότητες σε καιρούς κρίσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Διάβασα το έγγραφο αυτό θέσεων του Κοινοβουλίου και είναι πραγματικά εξαίρετο, οπότε θα περιοριστώ σε δύο σημεία μόνο. Πρώτα απ' όλα, στον τίτλο 2 που αφορά το Ταμείο Γάλακτος. Εκεί πέρα υπάρχει πρόταση να, πρόταση να συζητήσουμε προτάσεις για μόνιμο Ταμείο Γάλακτος. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσε η Επιτροπή μας ή και το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω ότι σκεφτόταν εδώ πέρα η συγκήτρια γιατί το Ταμείο Γάλακτος υποτίθεται ότι θα ίσχυε άπαξ. Δεύτερον, τίτλος 1. Εκεί πέρα πρέπει να είναι η βασική μας προτεραιότητα για τα περισσότερα μέτρα και προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να βγούμε από την ύφεση και να προγραμματίσουμε για το μέλλον. Νομίζω βρίσκονται σε αυτό τον τίτλο όπως πήγε τα προγράμματα πλαίσιο και τα διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία συνοχής. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω ένα παράδειγμα από τον τίτλο 1. Πράγματι καλωσορίζουμε αυτή την αύξηση 16,9 στον τίτλο 1β. Δεν ξέρω βεβαίως αν σε τελική ανάλυση ε, είναι αρκετό γιατί γνωρίζουμε πως ε, οι δαπάνε στην αρχή των προγραμμάτων είναι αργέ και μετά αυξάνονται. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν το 6,9% επαρκεί και θα πρέπει να ρωτήσουμε και τα άλλα θεσμικά όργανα εάν θεωρούν πως επαρκεί αυτό το ποσό και μήπως ε, εάν τελικά θα καταλήξουμε σε άλλον διορθωτικό προπολογισμό. Δεν πρέπει να περιμένουμε μετά διορθωτικό προπολογισμό. Πρέπει τώρα νομίζω να δούμε τι θα γίνει με τις ε, υποχρεώσεις σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Ο κ. Γενικό Διευθυντή έχει το λόγο για σχόλια και παρατηρήσεις Oui, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα που ετέθησαν προς την Κομισιόν. Καταρχήν το πρόγραμμα 2020. Θα ήθελα να σας δώσω ένα νούμερο. Το δείχνει πώς συνδέεται το πρόγραμμα αυτό με τον προπολογισμό. Ακόμα κι αν ο προπολογισμό δεν είναι ουσιαστικά το εργαλείο εφαρμογή αυτού του προγράμματος, το πεδίο του δηλαδή, είναι πολύ πιο ευρύ σε σχέση με τον κοινωτικό προπολογισμό. Και υπάρχουν επιπτώσει οι πολιτικές που εφαρμόζονται και στις χώρες μέλη. Ωστόσο, επισημαίνω ότι για την Ευρώπη 2020 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι περίπου 58 δις δηλαδή περίπου το 41% του προϋπολογισμού της Ένωσης, δίνεται με τον α ή το β τρόπο προς το στόχο 2020. Και επιμέρους για να ληφθούν υπόψη ορισμένα αιτήματα της Κομισιόν γίνονται ορισμένοι νέοι επαναπροσανατολισμοί. Δεύτερο, για τους νέους. Που είναι ένα θέμα που όπως και η συγγήτρια και η Κομισιόν το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Δεν θα πρέπει να δούμε μόνο την α ή τη β γραμμή του προπολογισμού. Όπως τον τίτλο υπάρχει η νότης ενδράση ή κάτι άλλο παρόμοιο. Ο προπολογισμό πάει στους νέους είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε cross-cutting, δηλαδή αφορά πολλά σημεία. Υπάρχει σε πολλές γραμμές του προπολογισμού. Και αν δούμε τα νούμερα, το διαθέσιμα, αν Απάντως τι γραμμές που δεν αφορούν μόνο την νεότητα, που αυξάνονται. Όχι πάρα πολύ, αλλά αυξάνονται. Αν δω λοιπόν τα νούμερα Youth on the Move το flagship 2 του προγράμματος 2020 αυτό που γίνεται για τις διάφορες πηγές κινητικότητα έρευνους μούντους, έρασμους για ε, νέες ε, επιχειρήσεις people μεταξύ του 2010 και του 2011 έχουμε αύξηση 1,780 δις από 1,780 σε πάνω από 2 δηλαδή αύξηση 13,4% των κονδυλίων 13,4% για τους νέους με διάφορες πολιτικές της Ένωσης. Με ειλικρίνη λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται υπέρ των νέων στον προϋπολογισμό είναι σημαντική. πιλωτικά προγράμματα και πιλωτικές δράσεις. Θα περιμένουμε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο πριν την πρώτη ανάγνωση. Άκουσα τα σχόλια της κυρίας Γκρέσλε για τις εξωτερικές σχέσεις. τα ερωτήματά της και τα σχόλιά της για την αύξηση των διαφόρων θέσεων. Ο τίτλος 3 ήταν ένας από τους πολλούς που θυσιάστηκαν στις διαπραγματεύσεις του 2005 και γίνεται τώρα μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό προς το τέλος της χρονικής αυτής περίοδου. Αλλά τονίζω ότι τα νούμερα στον προϋπολογισμό ανταποκρίνονται ακριβώς στον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Δεν υπάρχει τίποτα που να εκπλήσει όσον αφορά την εξέλιξη στα νούμερα αυτά. Τέλος, θα επανέλθω στην παρατήρηση της εισηγήτριας για την παράγραφο 56 διευκρινίζω ότι και εμείς έτσι ερμηνεύουμε το κείμενο. Η αύξηση του διοικητικού προπολογισμού της Κομισιόν είναι 2,9% που σημαίνει ότι το μερίδιό της στον διοικητικό προπολογισμό μειώθηκε σε σχέση με τα άλλα όργανα. Μπορεί εσείς να ερμηνεύετε διαφορετικά το κείμενο ανάλογα με το πώς έχει συνταχθεί και τι θα επικρατήσει τελικά ως <clears throat> κείμενο. Γενικά λοιπόν, από τη μεριά της Κομισιόν, ακούσαμε αυτά που υπόθηκαν για τον προπολογισμό, που δεν είναι ένας προπολογισμός post-crisis, είναι ένας προπολογισμός που έρχεται ακριβώς στο μέσο μιας κρίσης. Όταν συντάχθηκε ήταν ένας προπερισμός post-crisis, μετά την κρίση. Αλλά δεδομένου των προγραμματισμών, με τον τρόπο που κινούνται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να παίξουμε κάπως με τον αφιτοβήτα τρόπο τον προπολογισμό αυτό. Το κάναμε πέρυσι με το πρόγραμμα ανάκαψης Πάντως, σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και βρισκόμαστε σε κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Θα έχει επίπτωση στον προπολογισμό της Ένωσης η κατάσταση αυτή. Σας θυμίζω όμως ότι η διάρθρωση του κοινοτικού προπολογισμού είναι πολύ διαφορετική από τη διάρθρωση των εθνικών προπολογισμών. Και το τι περιθώρια λιγμών μπορούμε να έχουμε εμείς μπορεί να έχει μερικές φορές αρνητικό αντίκτυπο στις συνθήκες ανάκαμψης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί και συνετοί όταν πάμε να προσαρμόσουμε τον προπλησμό της Ένωσης προς τη ΒΑΤ Α ή τη Β κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε και Διευθυντά. Να κάνω κι εγώ μερικά σχόλια πριν η Συντόνια πάρει το λόγο για να κλείσουμε το σημαντικό αυτό σημείο. Όπως μας είπε ο κύριος Ζουανζόν, εδώ και μερικές εβδομάδες ζούμε μια νέα σημαντική κρίση, τρίτη θύελα, που δεν είχε προβλεφθεί όταν συντασσόταν αυτό το σχέδιο προπολογισμού. Σε 18 μήνες ο κόσμος στην Ευρώπη έζησε τρεις μεγάλες θύελες. Πρώτη, η χρηματοπιστωτική, η κρίση του ιδιωτικού χρέους μερικές μεγάλες τράπεζες σε όλες τις χώρες βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Δεύτερη θύελα, συνέπεια της πρώτης, η πρώτη σοβαρή ύφεση μετά τον πόλεμο. Οικονομική θύελα, που δυστυχώς έπληξε όλες τις οικονομίες μας και έμεσα και τους εθνικούς προπολογισμούς. Εδώ και κάμπους μήνες. Και εδώ προσθέθηκε μια τρίτη θύελα, καταγίδα, η κρίση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη. Αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγκάστηκε να υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι διότι η διεθνής οικονομική παίκτες κατά κάποιο τρόπο άρχισαν να διερωτώνται αν αγοράσαμε ορισμένες κρατικές ομολογίες ή ομόλογα μάλλον τίτλους που είναι αυτό που λέμε sovereign debt, κρατικό χρέος μήπως αγοράζουμε εξίσου τοξικά παράγωγα όπως ήταν τα subprimes στα αμερικάνικα πριν από 18 μήνες. Εκεί είχαμε φτάσει. Τρίτη φιέλα αυτή. Σήμερα δεν ξέρουμε σε ποια, ποια θα είναι η κατάσταση των οικονομιών μας μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες. Δεν έχουμε ορατότητα ως προς το ποιες θα είναι οι πραγματικές ανάγκες για τους προπολογισμού. Πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτής της κατάστασης. Φυσικά δεν κατηγορούμε την Κομισιόν που δεν πρόβλεψε αυτή τη θύελα. Εδώ και μια εβδομάδα κανένας από εμάς δεν την είχε προβλέψει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως. Λάβουμε υπόψη τις δύο πρώτες θύελες στους προπολογισμούς 2008-2010 με το Ευρωπαϊκό Μερίδιο, το πρόγραμμα δράση, ε, ανάκαμψης όπως υπόθηκε. Τώρα θα πρέπει να αγγιθεί υπόψη και αυτή η νέα τρίτη κρίση. Φυσικά όλοι έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το 2011 θα εφαρμοστεί η νέα δημοσιονομική διαδικασία που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ο Γκέραν Φέρμ σωστά τόνισε την ανάγκη να ορίσουμε προτεραιότητες στον τριμερή διάλογο. Τακτική αυτό για μας, επιλογή. Θα κάνουμε μια shopping list όπως πάμε να ψωνίσουμε στα μαγαζιά τα Χριστούγεννα ή θα είμαστε σε θέση να πούμε για μας υπάρχουν δύο ή μία ή τρεις ή τέσσερις προτεραιότητες μόνο, μόνο. Ζούμε μια έκτακτη κατάσταση, το Κοινοβούλιο επιμένει σε ένα σημείο μόνο, ενδεχομένω. Το μεγάλο πολιτικό ερώτημα έναντι των κρατών μελών είναι ενώ δεν έχουμε αλλάξει το σύστημα των πόρων που τροφοδοτούν τον κοινωνικό προπολογισμό, είναι το εξής πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να δεχτούν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στον ευρωπαϊκό προπολογισμό το 11 με βάση τη σημερινή συγκυρία. Μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει. Ταυτόχρονα όμως οι χώρες που υποχρεώθηκαν να, να αυξήσουν το έλλειμμα και το χρέος τους για να βοηθήσουν τις χώρες που, μέλη που ζουν δυσκολίες και αυτές θα διστάσουν να το κάνουν. Εμείς, Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, ενώ παράλληλα δίνουμε μαθήματα στα κράτη-μέλη λέγοντας ότι τα δημόσια νομικά τα κακοδιαχειριστήκατε, θα έχουμε μεγάλη δυσκολία να εξηγήσουμε ότι πρέπει όλοι οι άλλοι προπολογισμοί να μειωθούν, αλλά ο δικός μας να αυξηθεί. Και δεν λαμβάνουμε υπόψη με αυτές τις τρεις κρίσεις στην πραγματικότητα τα περισσότερα κράτη-μέγη της Ένωσης ζουν πάνω από τα μέσα που διαθέτουν. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ο τρόπος να επαναφέρουμε το βιωτικό μας επίπεδο σε αυτό που είμαστε σε θέση να χρηματοδοτούμε. Ταυτόχρονα όλοι οι οικονομολόγοι αναγνωρίζουν ότι αν σε μια φάση ύφεση όπως αυτή που ζούμε σήμερα και βγαίνουμε με δυσκολία αν ε, ε, ε, μειωθούν παντού τα δημόσια οικονομικά, θα έχουμε ύφεση. Ένα φαύλο κύκλο ή μια προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου. Κάθε χώρα μα προσπαθεί να βρει λύση, ο καθένα μόνο του. Κατά τη γνώμη μου όμω, η νέα κρίση οφείλει να παροθήσει όλες τις χώρες μέλη να προσπαθήσουν να βγουν από την κρίση μαζί, όλοι μαζί. Μαζί βρήκανε μία λύση προς τα πάνω στην κρίση του δημόσιου χρέους που εκφράστηκε έντονα την περασμένη εβδομάδα, πιστεύω ότι θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρούνε από κοινού μια λύση, μια λύση πάλι έξοδος προς τα άνω, από μια δημοσιονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε όλοι μας. Χώρες που διαχειρίστηκαν καλά τα οικονομικά τους πριν την κρίση, που τα κάκο Και μια τελευταία παρατήρηση κυρίως προς την Κομισιόν. Αλλά έμεσα θα ακούσει και το Συμβούλιο και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι. Στο πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες υπάρχουν διατάξεις, όροι, που όσον αφορά τα νούμερα, τα πιο σημαντικά νούμερα, λένε ότι τα κράτη-μέλη στον εθνικό τους προπολογισμό δεσμεύονται να δανειστούν, να δανείσουν, να δώσουν εγγυήσει κλπ. Αυτό δεν μα αφορά άμεσα. Υπάρχει όμω και ένα όρο κάπου, με βάση το άρθρο 122 τη συνθήκη, όπου η Ένωση και αυτή μπορεί να δανειστεί και να δανείσει. Θα ήθελα να με επιβεβαιώσετε ότι ο μηχανισμός που θα ισχύσει, που θα συσταθεί και θα ισχύσει, ότι θα είμαστε διαφανή ειλικρινείς, αυστηρή ότι δεν θα δημιουργήσουμε εκτός προϋπολογισμού σημεία, εκτός προϋπολογισμού, ούτε με την έννοια τη δημοσιονομική, ούτε με την έννοια την πολιτική. Μη δημιουργήσουμε δηλαδή παράλληλα με τους επίσημους λογαριασμούς, και για μας είναι ο κοινωνικός προϋπολογισμός, αυτό, άλλα παράλληλα έγγραφα και διαδικασίες που θα υπάκουν σε άλλους κανόνες και που θα ήταν ένα είδος το κρυμμένο παγόβουνο, κρυμμένο τμήμα του παγόβουνου. Πριν από 18 μήνες είδαμε τι έγινε με μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες που ανάλαβαν τέτοιου είδους δεσμεύσεις εκτός προπολογισμού, εκτός ισολογισμού μάλλον. Δεν πρέπει εμείς να δώσουμε το κακό παράδειγμα. Εμείς η δημόσια αρχή δημιουργώντας τέτοια πράγματα εκτός προπολογισμού. Δεν ξέρω πώς λογιστικά, νομικά και πολιτικά τα κράτη το καθένα στη χώρα του θα διαχειριστούν το τμήμα που ο καθένας δίνει μέσω του εθνικού προπολογισμού στο πρόγραμμα σωτηρία του Σαββατοκύριακου, πάντω θα πρέπει να φροντίσουμε να επαγρυπνούμε γιατί η ευθύνη μα είναι το κοινοτικό κομμάτι αυτού του προγράμματος σωτηρίας αυστηρά να μην μπορεί να υποστεί κανενός είδους αρνητική κριτική, διότι έχουμε υποχρέωση έναντι του πολίτη όσον αφορά, τις, ε, όσον αφορά την εμπιστοσύνη όλων αυτών που παίρνουν μέρος στο οικονομικό σύστημα. Μετά από όλες αυτές τις παρατηρήσεις, η συγγετριά μας θα μας πει ό,τι έχει να μας πει για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας για εκείνου που <clears throat> τους άρεσε η έκθεση, πολλά ευχαριστώ θέλω να πω. Και για εκείνου που είχαν επικρίσεις ή ε, παρατηρήσεις και σε εκείνου μεγάλες ευχαριστίες. Προσβλέπω στο να δω τι ε, τροπολογίε σα φυσικά και μέχρι τις 12 Μαΐου το μεσημέρι έχουμε χρόνο ακόμα. Ξέρω δεν επαρκεί, δεν είναι αρκετός αυτός ο χρόνος, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τις προτάσεις σας με γραπτό κείμενο και θα προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη. Θα ήθελα, Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, να αναφερθώ σε κάποιες από τις παρατηρήσεις. Δεν θέλω να είναι καθοριστικές, τελεσίδικες αυτές οι παρατηρήσεις, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις. Βρισκόμαστε σε μια δραματικού χαρακτήρα κατάσταση. Εμεί τα μέλη τη Επιτροπή Προπολογισμών, φυσικά και όλοι οι πολιτικοί άνδρε και γυναίκε που εμπλεκόμαστε στα τεκτενόμενα βλέπουμε την κρίση, όλα αυτά τα θέματα από τι πρώτε σελίδε των εφημερίδων ήδη. Αυτά τα θέματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες είναι σαφές αυτό, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε και τα όρια αυτής της έκθεσης για τον προϋπολογισμό του 2011 συγκεκριμένα. Υπάρχει ανάγκη να θέσουμε κέντρα βάρου ε, μεγάλων διαστάσεων στην έκθεση, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε και πειθαρχημένοι και ρεαλιστικοί, ρεαλιστέ. Ε, αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια διαφορά, μεταξύ του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των προπολογισμών των κρατών μελών στα κρατη και αυτό, αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Και αυτό είναι το γιατί έχουμε και δυσκολίες να, να ανταποκριθούμε και να αντιδράσουμε στην κρίση. Και αυτό γιατί. Διότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί και φέτος και κάθε χρόνο έχουν ελλείμματα και μια, αρνητικό ισολογισμό. Αλλά <clears throat> στον ευρωπαϊκό προπολογισμό έχουμε πλεόνασμα και επιστρέφονται κονδύλια στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ουσιαστικότερη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πλασμάτων μεταξύ αυτών των δύο δημιουργημάτων μας στο επίπεδο του προϋπολογισμού και καμιά φορά είναι και δύσκολο να, να εξηγεί κανείς στους πολίτες πώς επιστρέφουμε κονδύλια στα κράτη-μέλη. Το κάνουμε αυτό κάθε φορά και ξαφνικά η κατάσταση βλέπετε ότι διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο και έχουμε ε, κονδύλια που ε, περισσεύουν. Όμως είναι ένα πολύ περιορισμένο μέσο ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκριθούμε στα προβλήματα των κρατών μελών. Μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούσαμε καθόλου τα κονδύλια του προπολογισμού όσον αφορά τα προβλήματα των κρατών μελών. Έχουμε το περιορισμένο μέσο αντιστάθμιση, balance facility για να εγγυόμαστε πιστώσει. Είναι περιορισμένη εμβέλεια σε αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε πρέπει να γίνει μια διαρθρωμένη σε βάθο συζήτηση συζήτηση μεταξύ της Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ίσως όμως θα ήταν, ίσως, πώς να το πω, πρόημο να, έχει, να είχε γίνει κάτι τέτοιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011. Τώρα, παρόλα αυτά, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Όχι για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στους εθνικούς του προπολογισμού Δεν είναι αυτή η δουλειά του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και αν θέλουμε να είναι αυτή η δουλειά του πρέπει σε βάθος να επανεξετάσουμε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο στοχεύουμε και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πούμε είναι ο συγκεκριμένος ρόλος να χρηματοδοτήσουμε εγχειρήματα που δεν μπορούν να ε, αντιμετωπιστούν ατομικά επιμέρους από τα κράτη-μέλη αλλά μέσα σε ένα ε, πλαίσιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητές μας. Γι' αυτό επέλεξα το θέμα της ε, νεολαίας, γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση, η διασυνοριακή, η διαμεθοριακή και της κινητικότητας. Αυτή η πρόσθετη αξία που αποκαλούμε ε, και μπορεί να δώσει αυτή την μεγάλη ουσιώδη διαφορά. Και μέσα στο πλαίσιο το συγκεκριμένο της ε, περιορισμένης εμβέλειας έκθεσής μου και αυτό αναφέρεται και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης. Δεν είμαι πάλι σίγουρη ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός το μέσο το εργαλείο για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Ας μην δεν έχουμε αυταπάτες. Αν δεν έχουμε νομοθετικές αλλαγές για να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά την πολιτική απασχόληση, δεν θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης με τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και αυτή η παρατήρηση αφορά και γενικότερα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά αυτή η συζήτηση ελπίζω ότι θα μπορέσει να δώσει ρυθμιστικά πλαίσια και νομοθετικά εργαλεία για να πετύχουμε αυτή τη στοχοθέτηση. Δεν είναι ότι ε, δεν είμαι φάνταστη για να εντάξω πολλά θέματα μέσα αυτήν την έκθεση, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για τα θέματα αυτή τη έκθεση. Τώρα, για το 2011, τον προπολογισμό και τι παρατηρήσει σα εξειδικευμένοι εισηγητέ και ε, οι εξειδικευμένε επιμέρους κοινοβουλευτικέ επιτροπές και συνεργασία με αυτούς και αυτές. Στο μέτρο του εφικτού, μέσα σε αυτό το πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα, Συνεργάζομαι με κοινοβουλευτικέ επιτροπέ ε, όσον αφορά του ε, επιμέρου εισηγητέ. Είχα μια συνάντηση μαζί του. Είχα επίση ε, ενημερώσει με ηλεκτρονικά μηνύματα emails όσον αφορά και το χρονοδιάγραμμα και τα εργαλεία, τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, ενθαρρύνοντά του να καταθέσουν και τροπολογίε και σε σχέση με θέματα για τη γνωμοδότηση από πλευρά του. Γνωρίζω ότι υπάρχει πίεση χρονική το πλαίσιο τη οποία εργάζονται. Στις, ε, με τους εισηγητές ε, θα ε, συνέρθω στις 19 Μαΐου πρωτού ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Ελπίζω ότι θα υπάρχει μια δυνατότητα έτσι στο χρόνο να συζητήσω μαζί τους τροπολογίες που θα μπορέσουν να κατατεθούν. Από πλευρά μου υπάρχει κάθε προθυμία να συμπεριλάβω τις δικές τους παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους ακόμα και μέσα σε αυτό το πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Μια άλλη τώρα παρατήρηση που αφορά θα έλεγα ναι, πρέπει να ανταποκριθώ σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντή όσον αφορά το πρόγραμμα για την, τους, τους νέους. Για τα κονδύλια για τους νέους δεν είναι μια δική μου προσωπική ατομική αιμονή, όχι δηλαδή ότι ε, σε σχέση με το να αναφέρετε το θέμα ε, των ε, νέων και να θέλω να καλύπτεται κάτι υποχρεωτικά. Το θέμα της ε, εκπαίδευσης, κατάτησης με μεγάλη ποικιλία πολλών κονδυλίων που εμπλέκονται και έχουμε και σε σχέση με την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση συγκεκριμένα ερωτήματα και πιστέψτε με, καλύπτεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το θέμα αυτό, αλλά δεν μπόρεσε να μου δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς τα στοιχεία ποιοι είναι οι αποδέκτες νέοι ή ποιοι άλλοι. Κανείς δεν έχει, ας το πω έτσι, εξειδικευμένη εικόνα των εποφελούμενων όσον αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση, την ηλικία τους των αποδεκτών και ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά εργασίας για αυτούς. Πράγμα το οποίο είναι προβληματικό. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτών των κονδυλίων και τι γίνεται με αυτά τα λεφτά. Επίσης, γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα προγράμματα υποδημοσιονομική πτυχή πιστεύω ότι είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικά και έχω θέσει ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένω απαντήσεις με υπολογισμού όσον αφορά το Youth in Action και το Lifelong Learning, ιδιαίτερα Youth in Action, σε σχέση με την εκτέλεση δραστηριοτήτων, κάλυψη δραστηριοτήτων για τους νέους, non-school skills, δηλαδή παροχή δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ξένες γλώσσες, ε, γνώσεις, ε, ε, εξωσχολικών τέτοιων δραστηριοτήτων, αν υπολογίσετε ποιο είναι το κόστος αναϋποθελούμενο για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων για τους νέους. Αν χρηματοδοτείτε, για παράδειγμα, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα εκπλαγείτε. Είναι πανάκριβα τα μέτρα αυτά αν, το, αν τα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και αν τα αναλάβει το Youth in Action είναι πολύ φθηνότερα. Εκπληκτικό αυτό το συμπέρασμα. Αναμένω να μου δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συμπεράσματά της, τα στοιχεία της, να δούμε σε τι καταλήγουν. Είναι θέμα, αν θέλετε, ιεράρχησης πολιτικών προτεραιοτήτων. Επίσης, αποτελεσματικότητα των κονδυλίων που έχουμε στη διάθεσή μας στη χρήση τους. Θέλω να κατανοήσετε επίσης ε, τους βαθύτερους λόγους για αυτή την τοποθέτησή μου και άποψη που έχω. Και είναι ένας τρόπος να αυξήσουμε την εμπλοκή των πολιτών μας. Όχι μόνο να παρέχουμε υπηρεσίες, αλλά να προσκαλέσουμε και να οδηγήσουμε στο να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι πολίτες και να εμπλέκονται περισσότερο. Υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο σε όλα αυτά, βλέπετε. Θα ήθελα να απαντήσω και να ανταποκριθώ σε ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε όσον αφορά το Ταμείο Γάλακτος για τα σχολεία. Αυτή ήταν η αρχική επιθυμία της Ευρωβουλής. Ε, να εξετάσουμε μια, ένα μόνιμο πλαίσιο μόνιμης ρύθμισης ή λύσης. Αυτό που λέω στην έκθεσή μου είναι ότι θα ήθελα να δω την αξιολόγηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν επιτυχέ το εγχείρημα ή όχι όσον αφορά το Ταμείο Γάλακτο. Μάθαμε κάτι. Τι είναι αυτό που μάθαμε και πώς λειτουργεί. Και αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε ή όχι αυτό το πρόγραμμα. Δεν έχουμε ακόμα αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά. Είναι λοιπόν κάτι που είναι έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα ώστε να το ικανοποιήσει και να <clears throat> ακολουθήσει αυτή η αξιολόγηση των ε, δράσεων του Ταμείου Γάλακτος. Αυτή λοιπόν όλη η προσέγγιση της Ευρώπης 2020, αυτή η νέα ονομασία των υφιστάμενων προγραμμάτων. Είναι κάτι που πρέπει να τελούμε ενεγρηγόρση, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δούμε είναι κάποιο, δίνει κάποιο αποτέλεσμα σε σχέση με τη νέα ονοματολογία, σε σχέση με τη συνεισφορά στην Ευρώπη, τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 ή όχι. Είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, λαμβάνοντας υπόψη και κάποιους κινδύνους που υφίστανται, γιατί μπορεί να υπάρχει και σύγχυση όσον αφορά την ονοματολογία για κάποια, α το πω έτσι, ονόματα τα οποία για μας αντικατοπτρίζουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ένα προϊόν το οποίο έχει συγκεκριμένο όνομα. Όταν αυτά α, αλλάζουν ονοματολογία και ονομασία, τότε δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και πρέπει να δούμε ποια είναι η συνεισφορά τους στην Ευρώπη 2020. Μια αφετηρία, στο το πω έτσι, μια εκκίνηση συζήτησης αυτών των θεμάτων. Αν ξέχασα κάτι, να με συγχωρέσετε. Σημείωσε και κοιτάζω να δω αν έχω ξεχάσει κάτι και απομένει κάτι να σας αναφέρω. Όπως σας είπα αναμένω οπωσδήποτε τις τροπολογίες σας και θα τις εξετάσω και θα προσπαθήσω να τις συμπεριλάβω στο μέτρο του εφικτού και να ανταποκριθώ όσο γίνεται. Ένα σημαντικό θέμα τώρα που αφορά, <clears throat> ας το πω έτσι, την ε, έκθεσή μου. Δεν, είμαι, δεν αισθάνομαι πάρα πολύ ε, άνετα συζητώντας τα θέματα της εντολής μέσα σε αυτή τη διατύπωση, σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε εδώ μπροστά μας. Πιστεύω αυτά τα σημεία, παρότι είναι πάρα πολλά, είναι μια αφετηρία για μας, μια κίνηση για να <clears throat> μπορέσουμε να συγκλίνουμε και να εμβαθύνουμε. Δεν θέλω κάτι να αποκλείσω σε αυτή τη φάση, αλλά είμαι, θα έλεγα, σίγουρα πρόθυμη να εξετάσω σε μεγαλύτερο βάθος, σε, με μικρότερο αριθμό τέτοιων προτάσεων. Σε ένα, ας το πω έτσι, στενότερο πλαίσιο στοχοθέτησης, να συζητήσουμε κάποια από τα ουσιώδη στοιχεία για την εντολή μας. Και σίγουρα είμαι πρόθυμη να υποβάλω και κάποιες προτάσεις και ιδέες για το, το πλαίσιο της εντολής. Αλλά πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και να το συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε συντόνια και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος σε αυτόν τον ενδιαφέροντα γύρο. Σας θυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μεθαύριο, 12 του μηνό 12 η ώρα. Δεύτερη συνεδρίαση τη ομάδα εργασίας με του εισηγητέ των άλλων επιτροπών προβλέπεται για τις 19 Μαΐου. Προθεσμία τροπολογιών θα έχει περάσει βέβαια, αλλά όπως είπε ο συνάδελφος Φέρμα, να είμαστε σε διεθνή επαφή με τις άλλες επιτροπές. Πάντως το input των άλλων επιτροπών θα είναι σημαντικό όταν θα έρθουν οι καθ' αυτό στον προπολογισμό. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 2 Ιουνίου. Ολομέλεια μάλλον 15 ή 16 Ιουνίου. Και ο τριμερής διάλογος 30 Ιουνίου. Μέχρι τότε θα πρέπει να βρούμε μια λύση προκειμένου να βρούμε μια, ένα συμβασμό μεταξύ μας στο τι θεωρούμε ότι έχει προτεραιότητα. Θα το βάλουμε σε μια συνεδρίαση των συντονιστών και μετά να το συζητήσουμε και κλεισμένο το θεωρώ ενδεχομένω σε συνεδρίαση τη Επιτροπή. Α συνεχίσουμε. Μα πήρε λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι προβλέπαμε το σημείο αυτό. Ας πάμε λίγο πιο γρήγορα με τα υπόλοιπα. 5. Διορθωτικός προπολογισμό αριθμός 2. Κοινωνική Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Περιφερειών. Νέα στοιχεία δεν έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Manca va nous donner son l'état de du débat sur ce sujet. Ο κύριος Μάνκα θα μας πει τι γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γι' αυτό το θέμα για το διορθωτικό προϋπολογισμό δεν έχω τίποτα καινούργιο από την τελευταία μας συνάντηση. Αναμένουμε τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Εξίσου αναμένουμε το όπως και για αυτή τη γνωμοδότηση αναμένουμε τη γνωμοδότηση για το τμήμα για το κοινοβούλιο. Επίσης και λόγω των διαφορετικών απόψεων, των απόψεων των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών με θετική τοποθέτηση ή προσέγγιση και οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν περισσότερες αρμοδιότητες και πολύ περισσότερη δουλειά και επιβάρυνση από αυτή τη δουλειά, βάρος από αυτή τη δουλειά με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας 10,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι το ποσό. Και παρότι τον Απρίλιο στην Ολομέλεια ήδη πώς να το πω, είχαμε τον διορθωτικό προϋπολογισμό επί του οποίου συζητήσαμε και συμφωνήσαμε, μπορεί αυτό το ποσό να μειωθεί τελικά, διότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές δεν θα είναι σε θέση να ε, εκμεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το ποσό πλήρως. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στη δική σας έκθεση όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα, την, ε, ε, διαδικασίες ε, με, με βάση τις συνθήκες της αγώνας. Εδώ στο σημείο 13 αναφέρεται η διαπίστωση ότι στη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων θέλουμε να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία στις διάφορες φάσεις ε, της ε, δημοσιονομικής διεργασίας στην εξέταση θεμάτων προϋπολογισμού. Όμως, μια και εδώ και δύο μήνες δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν το Συμβούλιο έχει άλλη άποψη ή όχι. Και μια και εμείς εξαρτώμαστε από αυτό, θα έπρεπε να προστείλουμε ένα μήνυμα ήδη σήμερα ότι χρειαζόμαστε αυτόν τον τριμερή διάλογο. Πρέπει να διεξαχθεί. Και ένας τριμερής διάλογος που ε, στις 30 ε, Ιουνίου θα διεξαχθεί, διεξάγεται σε μια σχετικά, θα έλεγα, όψιμη ε, ιστερότερη χρονική στιγμή. Αυτά ήθελα να πω και να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ και θα πρότεινα να μην αναλώσουμε ιδιαίτερα πολύ χρόνο για αυτό το σημείο ή μάλιστα και για τα δύο σημεία της ημερησίας διάταξης 5 και 6 τηρήσαμε μέχρι τώρα το χρονοδιάγραμμά μας και όσον αφορά τον διορθωτικό προϋπολογισμό τμήμα Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, εγκρίναμε ή προχωρήσαμε ε, χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας ε, την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής, όμως προχωρήσαμε και αναμένουμε να υποβληθεί η άποψή τους ιστερότερα. Ταυτόχρονα ξεκινούν συζητήσεις μεταξύ της Ισπανικής Προεδρίας και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ευρωβουλή. Εμείς όμως ως Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουμε τον ρόλο μας που τον υλοποιήσαμε και τις αρμοδιότητες μας και ανταποκριθήκαμε σε αυτές. Θα δούμε με τους συντονιστές ε, πώς, ε, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε ώστε να μπορέσουμε το δυνατόν πιο γοργά να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και ελπίζουμε με την σύντομη υλοποίηση ενός ε, τριμερούς διαλόγου όπως ανέφερε και ο εισηγητής. Περνάμε λοιπόν στη συνέχεια στο σημείο 7. Ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2007-2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Απριλίου ενέκρινε μια έκθεση για την αξιολόγηση αξιολόγηση της λειτουργίας της ε, διοργανικής συμφωνίας. Αυτή η έκθεση έχει υποβληθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μπέγκε να μας πει ποια είναι η άποψή του σε σχέση με αυτά τα θέματα. Και ίσως ε, εν παρόδο θα μπορούσε να αναφερθεί και στο σημείο 8, τεχνικές προσαρμογές του δημοσιονομικού πλαισίου. Ράιμερ, έχει τον λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά το σημείο 8 βασίζεται στα σημεία 16 και 17 της διοργανικής ε, συμφωνίας και μιλάμε ε, κυρίως για τεχνικές προσαρμογές που πρέπει να κάνει η Κομισιόν και θα ήθελα να μας πει και κάποια πράγματα η Κομισιόν. Κυρίως μιλάμε για αποκλήσεις ε, του ΑΕΠ, κυρίως τρία κράτη-μέλη σε κάτι το οποίο βεβαίως θα έχει αλλαγές σε σχέση με την πολιτική συνοχή για αυτά τα τρία κρατημέλη. Τώρα όσον αφορά την έκθεση Κομισιόν για την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου θα ήθελα να κάνω πρώτα απ' όλα τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα με αυτά τα οποία λέγονται επί της αρχής είμαι αρκετά ικανοποιημένος γιατί το εύρος ε, των προβλημάτων εφαρμογής που είχαμε τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζεται ικανοποιητικά. Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος όσον αφορά βεβαίως τα πολιτικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν αυτό βεβαίως, ε, εντάξει, παρακολουθείτε η κατάσταση, αλλά το τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εφαρμογή και τις ε, τυχόν βελτιώσεις, ε, νομίζω αυτό γίνεται με βάση την αξιολόγηση που κάνει η Κομισιόν και γράφει εκεί πέρα στο τέλος του εγγράφου πως θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις σύμφωνα με τις επιλογές που έχουμε μόλις ε, ξεκαθαριστεί το τι επίδραση θα έχουν αυτές στον προπολογισμό. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν από την Κομισιόν. Είναι διατεθειμένη να συμπεριληφθούν ε, τμήματα αυτής της συζήτησης, της αναγκαίες πολιτικές προσαρμογές που θα υπάρξουν ε, με βασική την εφαρμογή του MFF και του EV, γιατί δεν ε, ξέρω πώς θα μπορούμε να περιμένουμε για όλα αυτά τα ζητήματα μέχρι το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις ανάλογες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Και να σας πω κάτι ήδη από τώρα, ε, κάτι το οποίο πραγματικά με τρομάζει. Θεμητό και σωστό, εντάξει τώρα ξεκινάω από το τέλος λίγο, η Κομισιόν να λέει στα προβλήματα των περιθωρίων τα οποία συνεχώς μικραίνουν και εξαφανίζονται να εξετάσει τυχόν επιλογές για την χρηματοδότηση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων είτε μιλάμε για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 είτε μιλάμε για τις συνέπειες των τομέα της ε, της κλιματικής αλλαγής ε, και πολλά άλλα και Μιλάει βεβαίως για το ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές παραδοσιακά, το τι δυνατότητες έχουμε με μετατοπίσεις, με το να υπάρξει το παραδοσιακό μέσο ευελιξίας, με το τι θα σημαίνει αυτό βεβαίως με τη μείωση του και την αύξηση του άλλου, ή να υπάρξει μια συνολική άνοδο συνολικού ορίου από το 2007 μέχρι το 2013 και μετά έχουμε μια άλλη προβληματική πρόταση. Λοιπές ε, δυνατότητες χρηματοδότησης όπως παραδείγματο χάρη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη ή δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν επίσης να εξεταστούν. Εντάξει, εγώ είμαι πάντα υπέρ του να αναζητούμε εναλλακτικέ λύσει ε, είτε στο πλαίσιο έτσι μιας εξέταση ιδεών, ε, εναλλακτικών λύσεων και να τι αξιολογήσουμε πολιτικά, να δούμε το τι μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί βεβαίω θα πρέπει να καταλήξουμε και σε κάποιους ε, συμβασμούς, αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις θεωρητικές εδώ πέρα δυνατότητες, λείπει κάτι, μια αναγνώριση της Κομισιόν, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει. Εντάξει, υπάρχουν τα προβλήματα της κρίσης κτλ. Και υπάρχει η δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουν τα κράτη-μέλη. Ναι, εντάξει. Ε, εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού, θεωρώ πως είναι κάτι εξαιρετικά το επικίνδυνο να μιλάμε. Τι θα κάνουμε στο μέλλον με τα άρθρα 310 και 311 της ε, συνθήκης που λέει πως όλα τα έξοδα και τα έξοδα της ε, κοινότητας ε, αναφέρονται, υπολογίζονται κατ' και αναφέρονται στον προπολογισμό της κοινότητας, 310. Άρθρο 3.11. Θα πρέπει η Ένωση να επιτυγχάνει τους στόχους της με τα διαθέσιμα μέσα. Αυτά δεν κολλάνε εδώ πέρα. Η Κομισιόν δεν ξέρω ποια πολιτική στάση τηρεί, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο ε, μήνυμα αυτό το οποίο στέλνει στο Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την Κομισιόν, τον Επίτροπο, να το διευκρινίσει αυτό εδώ πέρα, γιατί νομίζω πως αντιβαίνει με αυτά τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 3.10 και 3.11. Και απομακρυνόμαστε βεβαίω ακόμη περισσότερο από την κοινοτική μέθοδο. Γνωρίζω βεβαίως πως δεν είναι απλό λόγω των καθυστερήσεων που όλοι γνωρίζουμε να γίνουν οι δημοσιονομικές εκτιμήσεις εγκαίρως για το ποιες συνέπειες μετά θα έχουν στον προϋπολογισμό η συνθήκη, θα έχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Λέει η Κομισιόν πως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τα νομοθετήματα και μετά να δούμε ε, ποια θα είναι αυτή η δημοσιονομική αξιολόγηση. Ναι, αλλά Για το όνομα του Θεού δηλαδή, τα έχουμε συζητήσει και με τους ε, συντονιστές, κοιτά εδώ πέρα και τον κύριο Γκολτιέρη. Ε, λέμε εδώ πέρα πώς θα έχουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικών χωρίς μια διοργανική συμφωνία η οποία θα μιλήσει, θα αναφέρει βεβαίως και τον τρόπο λειτουργίας αλλά και ακριβώς τις δημοσιονομικές συνέπειες με βάση τις νέες αυτές δομές εργασίας. Δηλαδή αν δεν συνεννοηθούμε για το πώς θα πληρώνουμε και θα έχουμε και ένα μισοπρόθεσμο προγραμματισμό για τα επόμενα τρία χρόνια, ε, δεν υπάρχει καμία λογική και ο χρόνος πιέζει. Ε. Ή θα πρέπει να κάνουμε κάτι ή δεν ξέρω, τα επόμενα τρία χρόνια δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να βγούμε. Πρέπει να το πω αυτό εδώ πέρα ξεκάθαρα. Από την άλλη, η Κομισιόν όσον αφορά το ζήτημα της ε, εφαρμογής και ε, της χρήσης των ε, όρων παραγράφων της διοργανικής συμφωνίας λέει πως θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί εγκαίρως αλλά όσον αφορά τις τρέψεις διαδικασίες, ε, τις αναθεωρήσεις ε, από το Γαλιλαίο μέχρι το μέσο τροφίμων κτλ. Ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερο χρόνο για να βρει μία λύση και επανερχόμαστε στο ότι αφενός θα πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τον τρόπο λειτουργίας της Διοργανικής Συμφωνίας για να πούμε πως έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά όσον αφορά το τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τα ποσά, δεν βλέπουμε εδώ πέρα κανένα συσχετισμό. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει πιο... πώς θα ρεύσει καλύτερα αυτή η διαδικασία αν θέλετε. και να δούμε τι θα γίνει με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, πώς θα κινητοποιήσουμε τα ταμεία τα οποία έχουμε και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, το Ταμείο Αλληλεγγύης και το απόθεμα βοήθειας εκτάκτου ανάγκης και πώς θα κινητοποιηθούν όλα αυτά. Νομίζω είναι ε, όλα αυτά υπάγονται στο πώς θα προσαρμοστούμε στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, για να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Τώρα, εάν η Κομισιόν ε, μας λέει τι θα γίνει με την προσαρμογή στο MFF κτλ. Εδώ πέρα συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει. Μιλάει λοιπόν για την ευελιξία στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, αναφέρει λοιπόν πως υπάρχουν κάποιες προκλήσεις όπως η χρηματοδότηση του Κοσλοντούι, η χρηματοδότηση νέων εποπτικών αρχών, το μέσο μικροχρηματοδότησης, οι δραστηριότητες του GMIS, εδώ πέρα δεν ξέρω, θα ήθελα να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα και αυτά έχουν ληφθεί υπόψη, αλλά μετά μιλάτε για το έργο ITER και κάποια άλλα τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν στον προγραμματισμό έτσι ώστε τα διαθέσιμα περιθώρια τα οποία έχουμε σε πολύ σημαντικές ε, κατηγορίες ε, τίνουν σταδιακά προς το μηδέν. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, να μειωθεί δηλαδή η κατηγορία 2 και να ανεβούν, οι, μάλλον αυτό δεν θα είναι πλέον δυνατό τα επόμενα χρόνια, να μειωθεί η κατηγορία 2 για να αυξηθούν τα διαθέσιμα στις υπόλοιπες ε, κατηγορίες και να δούμε το πώς θα ε, συνεχιστεί αυτό το οποίο είχαμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Να σας υπενθυμίσω πως τον Ιανουάριο του 2005 στην αρχή των διαπραγματεύσεων με την Αυστριακή Προεδρία είχαμε παρουσιάσει ένα έγγραφο στο οποίο λέγαμε να ξέρουμε πως δεν είναι απλό να αλλάξουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά ως ηγετής είχα πει τότε πως πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 12 ε, δισεκατομμύρια πλέον για να μπορέσουμε να βγούμε. Και μου είπαν τότε πως τρελάθηκε ο εισηγητή του Κοινοβουλίου. Και σήμερα ήδη έχουμε φτάσει στα 8 δισεκατομμύρια στο ε, μισό του της διάρκειας αυτής της ε, περίοδου. Οπότε νομίζω πρέπει να εργαστούμε λίγο σοβαρά εδώ πέρα. Και η Κομισιόν αναφέρει πως οι κατηγορίες επίσης ένα α, κατηγορία 3 ε, και ειδικά 3β και η κατηγορία 4 έχουν σοβαρές δυσκολίες και πρέπει Νομίζω να υποθέτουμε πως ε, όσον αφορά όλο αυτό το πρόβλημα της ε, Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας θα έχει μία επίδραση στην κατηγορία 4 όπως και στην κατηγορία 5. Γιατί πολύ απλά αμφιβάλλω πως ε, θα καλυφθούν αυτά με το συνολικό πλαίσιο που υπάρχει. Μετά η Κομισιόν λέει πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε πως η δημιουργία της υπηρεσίας αυτής θα απαιτήσει περαιτέρω μέσα. Εδώ πέρα θα ήθελα να μας πούν κάποια πράγματα παραπάνω σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, εάν κάπου αλλού είχαμε μία περαιτέρω επιλογή. Θα μπορούσαμε ε, να δούμε τι θα γίνει και με την υπηρεσία εξωτερική δράση, αλλά πολύ απλά αυτό δεν συμβαίνει. Είπα λοιπόν λίγα πραγματάκια για τα διάφορα ταμεία. Τα αναλύει αρκετά λογικά η Κομισιόν, αλλά νομίζω πως αυτά τα πράγματα πηγαίνουν πέρα από την διοργανική συμφωνία. Πώς λειτουργεί δηλαδή η κινητοποίηση αυτών των ταμείων, τι γίνεται με τη χρηματοδότηση αυτών των ταμείων, να δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν αυτά τα ταμεία με την εντονότερη χρήση του Ταμείου της ε, παγκοσμιοποίησης, από πού θα προέρχονται σε μόνιμη βάση τα κονδύλια αυτού του Ταμείου και υπάρχει όπως σας είπα και το Ταμείο της ε, ε, αλληλεγγύης και των εκτάκτων, της εκτάκτης βοήθειας. Εντάξει, μιλήσαμε επίσης για την ευελιξία, το μέσο ευελιξίας. Φαίνεται πως ε, μας έδωσε περισσότερες δυνατότητες σε αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές από ό,τι στο παρελθόν, αλλά σωστά αναφέρει η Κομισιόν πως παραδείγματο χάρη το έτος 2010 το ποσό το διαθέσιμο είναι ήδη περιορισμένο στα 115 εκατομμύρια. Επιπλέον μιλάμε για το ότι υπάρχει μία νομοθετική ευελιξία, δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα εδώ πέρα για ένα 5% των ε, για ένα 5% απόκληση από τους πολιετής ε, φακέλους και αυτό νομίζω είναι ένα θέμα ε, για τις εξειδικευμένες επιτροπές του Κοινοβουλίου και όχι μόνο για την Επιτροπή Προϋπολογισμού ακριβώς ίσως για την μεσοπρόθεσμη αυτή αξιολόγηση των πολιετών προγραμμάτων. Θεωρώ πως ε, θα πρέπει να αναμένουμε από τις άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου όταν θα κάνουμε τα επόμενα βήματα της, ε, του πολιετούς προγραμματισμού να μας πει η κάθε επιτροπή και ίσως αυτό θα έπρεπε να το δούμε στην διαδικασία του 2011 να πούμε πως ε, το αργότερο το 2011 θα έχουμε μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση των πολιετών προγραμμάτων, γιατί αυτό απαιτείται και από την Κομισιόν, αλλά και από τις εξειδικευμένες επιτροπές, ε, δηλαδή που υπάρχουν οι προτεραιότητες, ε, που έχουμε μια προσέγγιση με την επικουρικότητα, που έχουν εξελιχθεί και που δεν έχουν διατεθεί τα υπάρχοντα μέσα αυτά αφορούν βεβαίως και τη σοβαρότητα του Κοινοβουλίου και πρέπει να τα δουν σοβαρά οι αρμόδιες ε, επιτροπές. Θα μπορούσε λοιπόν ε, και ο πρόεδρος να υπενθυμίσει εδώ πέρα ε, τις προθεσμίες αυτές στις άλλες επιτροπές, να υπενθυμίσει πως πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους εδώ πέρα για να υπάρχει και η απαραίτητη αξιοπιστία μας. Ενδιαφέρον είναι επίσης πως η Κομισιόν εδώ πέρα αναφέρει πως επειδή αυξάνεται λόγω των διαφέρων στόχων η ανάγκη χρηματοδότησης, πρέπει εδώ πέρα να υπάρξει και διάθεση από το μέσο ευελιξίας. Δηλαδή εδώ πέρα ομολογούμε πως έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και θα πρέπει να επιτευχθούν κάποια πράγματα τα επόμενα τρία χρόνια και αυτό πιθανώς δεν θα γίνει με το υπάρχον πλαίσιο ευελιξίας, το υπάρχον μέσο ευελιξίας. Εν τω μεταξύ, με την έγκριση του Συμβουλίου, δηλαδή με την διοργανική συμφωνία, λέμε πώς θα πρέπει να υπάρξει να αφήσουμε ένα περιθώριο σε όλες τις κατηγορίες. Δεν έχουμε ποτέ ορίσει πόσο μεγάλο θα πρέπει να είναι, αλλά παρόλα αυτά επειδή δεν γινόταν διαφορετικά με το πακέτο το οποίο φτιάξανε, φτιάξαμε καμία φορά φτάσαμε στο μηδέν με τη, με τη συμφωνία του Συμβουλίου γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Πώς θα ρυθμίσουμε αυτό το θέμα στο μέλλον, δηλαδή να υπάρχουν επαρκή περιθώρια ή τα έχουμε χρηματοδοτήσει όλα τόσο τσίμα τσίμα έτσι ώστε μέχρι το τέλος του πολιετούς ε, προγραμματισμού θα πρέπει να παραβούμε αυτά τα οποία γράφονται εδώ πέρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι έχει αναλύσει εδώ πέρα η Κομισιόν και να τα αναδιατυπώσουμε, να βγάλουμε τα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα, δηλαδή τι γίνεται με τα επαρκή περιθώρια που θα πρέπει να υπάρχουν. Ίσως θα έπρεπε να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό εντός των κατηγοριών, εντός των οροφών της κάθε κατηγορίας. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε όταν μιλάμε για την ε, διοργανική συμφωνία, για την διαδικασία του υπερπολογισμού και την αναθεώρηση, το ότι έχουμε ένα πρόβλημα με βάση των σημείων 22 και εξής στην ε, υφιστάμενη διοργανική συμφωνία πως ε, υπάρχει ένα όριο αναθεώρησης του είναι 0,03% του ΑΕΠ και ίσως θα έπρεπε να το επανεξετάσουμε, να το δούμε διαφορετικά από ό,τι κάναμε μέχρι στιγμής. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την ε, ισορροπία των ε, δημοσιονομικών αρχών, να μην το παραμερίσουμε δηλαδή αυτό το κομμάτι της ε, συνθήκης και να μην φτάσουμε, όπως σας είπα, το μέσο ευελιξίας να τίνει προς το μηδέν επειδή υπάρχει αυτή η ομοφωνία στο Συμβούλιο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ανταυτού και όσον αφορά τα τυχόν περιθώρια και όσον αφορά την αλλαγή του μέσου ευελιξίας αναφέροντας ίσως τα ε, ετήσια πλαφών στον προπολογισμό ή στα επιπλέον αποθεματικά που θα πρέπει να δημιουργηθούν. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν εδώ στην Επιτροπή μας και μετά να δούμε τις διαπραγματεύσεις για τη Οργανική Συμφωνία και να μην περιμένουμε τον επόμενο πολιετή προγραμματισμό. Αυτά έτσι γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, ως πρώτες ε, παρατηρήσεις. Πιστεύω πως ε, με βάση αυτή την έκθεση είναι σημαντικό πριν γίνει η συζήτηση για τα με προφορικές ερωτήσει στην Κομισιόν να δούμε αυτά τα σημεία για να μπορέσουμε να τα ενσωματώσουμε στην συζήτησή μας για να προετοιμάσουμε αυτή την έκθεση και μετά να δούμε ποιε θα είναι οι πολιτικές απαιτήσει που θα έχουμε ως Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τις αλλαγές της Λισαβόνας για το τι θα γίνει με αυτή τη ε, μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Αν Γένσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ρόιμερ. Πολύ καλή έκθεση αυτή της Κομισιόν. Μας δίνει μια σαφή εικόνα της κατάστασης και εξηγεί γιατί πρέπει να εξακολουθούμε να ασκούμε πίεση στην Κομισιόν για να μας κάνει μια αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως κάνουμε και με τη γραπτή ερώτηση. Τα περιθώρια είναι πολύ σφιχτά στην κατηγορία 1. Η Κομισιόν μας εξήγησε Υπάρχει ένα πρόγραμμα που στοιχίζει περίπου ένα δις και τα χρήματα δεν υπάρχουν να δούμε πού θα βρούμε τα λεφτά αυτά. Καλά, αυτό ήταν ένα. Με το Γαλιλαίο, τι γίνεται, μπορεί και αυτοί να χρειαστούν περισσότερα λεφτά. Υπάρχουν οργανισμοί που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ακόμη και όπου να είναι θα αρχίσουν να λειτουργούν. Πολλά πράγματα έρχονται. Έχουμε την κατηγορία 2, τα γεωργικά. Υπάρχουν χρήματα εκεί που κάθονται τα προηγούμενα χρόνια. Όχι τόσο πολύ τώρα πια. Υπάρχει διαφορά στις εκτιμήσεις αυτού εδώ του κειμένου και του προπολογισμού 2011. Ξέρω το, το πλεόνασμα μειώνεται. Και για το 2012 και 2013 ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το κόστος για τη γεωρική πολιτική δεν έχει χτυπήσει οροφή. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να το πιστεύει αυτό η Κομισιόν, πάντως έτσι βλέπουμε ότι θα έχουμε προβλήματα και στον τομέα αυτό. πρέπει να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Τα νέα αιτήματα από τη συνθήκη της Λισαβόνας, η εξωτερική υπηρεσία, δεν αναφέρεται όμως η πολιτική ή το διάστημα και άλλα που υπάρχουν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ξέρουμε ότι πολλά πράγματα έρχονται σε λίγο, έχουμε εξηγήσει, αλλά οι εξηγήσει δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επαρκέσουν όλα αυτά. Η Συντόνια πιο πριν είπε ότι ο προπολογισμό τη Ένωση είναι διαφορετικό από τον προπολογισμό των κρατών μελών. Δεν επιτρέπεται να έχει έγκλημα. Πρέπει να έχει πάντα πλεόνασμα. Η τεράστια διαφορά είναι ότι πέρα από, το γεωργικό προπολογισμό είναι ένα προπολογισμό για προγράμματα. Εφταετίως επί το πλήστον. Δεν υπάρχει μεγάλη ευελιξία. και τώρα έχουμε δέσει τα χέρια μας. Μην αφήνοντας επιπλέον περιθώρια. Ό,τι ιδέες και να έχουμε θα πρέπει να συνδεθούν με προγράμματα που έχουν ήδη αποφασιστεί ή εκτελούνται. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, τουλάχιστον να έχουμε ειλικρίνεια, να ξέρουμε πού πάμε. Γιατί είναι σαν να ξεγελάμε ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή. Λέγοντα ότι θα θέλουμε να εκτελεστούν ορισμένες πολιτικές ενώ δεν υπάρχει χρηματοδότηση γι' αυτό. Δεν δικαιολογείται. Πρόεδρε, ευχαριστούμε αν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το τρέχον, δείχνει ότι η μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός εθνικού προπολογισμού και του κοινοτικού είναι ότι ο εθνικός είναι για ένα έτος, ενώ ο κοινοτικός είναι για 7 χρόνια. Υπερβάλλοντας κάπως. Δηλαδή κάνουμε σαν να ψηφίζουμε έναν ετήσιο προπολογισμό, στην πραγματικότητα είναι παγωμένος για 7 χρόνια. Και αυτό δεν στέκεται ούτε τεχνικά ούτε πολιτικά πια. Γκέραντ Φέρμ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ράιμερ Μπέγκε. Συμφωνώ πάνω κάτω με την ανάλυση που μας έκανε. Και η έκθεση της Κομισιόν χρήσιμη είναι. Ανησυχώ όμω. Γιατί αυτό που λένε ότι υπάρχουν τρεις λύσεις χρησιμοποίηση το δημοσιονομικού εργαλείο η αναθεώρηση ή διαφορετική χρήση. Η άλλη αναθεώρηση αφορά μόνο το ίτερ και την αλλαγή του κλίματος. Αυτό παρά είναι παθητικό ως στάση. Στην έκθεση της Συντόνια υπάρχουν πολλές πολιτικές που δεν θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν αν δεν γίνει αναθεώρηση. Πέραν του ίτερ και της αλλαγής του κλίματος Πολύ παθητικό αυτό το συμπέρασμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί στο σημείο αυτό. Άσχετα με το ίτερ και την αλλαγή του κλίματος. Εκεί δεν έχουμε επιλογή. Επιβάλλεται. Επιβάλλονται αυτά στην αναθεώρηση. Αλλά πρέπει να το κάνουμε και για άλλα. Η Κομισιόν όμως δεν καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Το θέμα είναι τι κάνουμε με πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί θα είναι σημαντικό αυτό και για τον προπολισμό του 2011. Τι θα κάνουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αν η Κομισιόν μας ζητήσει μία πρόταση μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου, καλώς, αλλά αν δεν το κάνει, έχουμε την προφορική ερώτηση, αλλά μετά θα πρέπει πολύ σύντομα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πότε και πώς. Διαφορετικά θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Έλγα. Πιθανώς για να ξέρει αν ο δοντοτός τροχός της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα είναι πράσινος. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα, Πρόεδρε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή της και τον Ράιμερ Μπέγκε για το όσα μας εξέθεσε πιο πριν. Θα προσπαθήσω τις αντικρουόμενες αυτές απόψεις όσον αφορά τους στόχους να αναφέρω. Μία αναθεώρηση ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι αναγκαία όταν αφενός θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τις νέες προτεραιότητες και εκκινώντας από την κρίση και τις νέες απαιτήσεις, κλίμα, κλιματικές αλλαγές, νέα ανάπτυξη, νέες θέσεις απασχόλησης, νέα υλικά, καταπολέμησης ανεργίας των νέων, όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Αν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε πρέπει αυτό να κάνουμε. Με τη σημερινή δομή του προϋπολογισμού δεν γίνεται αυτό. <clears throat> Δεν θα είχαμε όλες αυτές τις αλλαγές ε, που έχουμε συζητήσει για μεταθέσεις και μεταφορές ε, κονδυλίων από το, από το Συμβούλιο. Με όλες τις διαφορές που έχουμε κομματικά όμως αυτό ήταν κοινό σημείο μεταξύ μας, ότι χρειαζόμαστε αυτή την αναθεώρηση για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε νέες προτεραιότητες. Ποιο είναι το ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή λοιπόν. Είναι αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε χρέη. Είναι σημαντικό και σωστό. Και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι και πολύ περιορισμένος. Όμως με κάποιο βαθμό η ελαστικότητα, αν τα τελευταία χρόνια την πετύχαμε, ήταν δυνατόν τα κράτη-μέλη να δίνουν νοπό χρήμα και στο τέλος τέλος αυτό με νέα δάνεια ή δανειοδοτικές ε, πράξεις χρηματοδοτήθηκε από τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο ο Αλέν Λαμασούρ είπε πιο πριν, ότι κατά κάποιον τρόπο τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες ζούσαμε πάνω από τις ε, δυνατότητές μας. Όλο περισσότερο χρεωνόμαστε για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Τώρα όμως στη Γερμανία με το 2011 δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πια με αυτή την πολιτική, διότι Πρέπει να σταματήσουμε να υπερχρεωνόμαστε. Πατάμε, τραβάμε το φρένο όσον αφορά την υπερχρέωση. Δεν είναι δυνατό λοιπόν με δάνεια να χρηματοδοτούμε αυτέ τι δράσει. Αυτό θα έχει και είναι αναγκαστικό επιπτώσει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η προθυμία τη Γερμανία και άλλων κρατών μελών να διαθέτουν περισσότερα κονδύλια στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, πράγμα το οποίο είναι συνέπεια από τις κοινέ μας αποφάσεις, Γαλιλαίο και όλα τα άλλα κοινά προγράμματα, αυτό θα σήμαινε με το πολύ μικρό περιθώριο που έχουμε και με τις νέες προτεραιότητες που έχουμε να χρηματοδοτήσουμε, ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση κονδυλίων του προϋπολογισμού. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ε, ότι όλα τα άλλα μπορεί να, ε, παρότι είναι ευκταία, να δούμε είναι ρεαλιστικά. Τι απορρέει από όλα αυτά. Αφενός ε, υπάρχει η δυνατότητα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αν δεν υπάρχουν νέα κονδύλια, να υπάρξουν μεταθέσεις, μεταφορές κονδυλίων. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επώδυνο, οδυνηρό, διότι πολλά από αυτά που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και με βάση τις αποφάσεις που έχουμε λάβει θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε, δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε και πρέπει να μετατεθούν. Η άλλη στρατηγική ή ο στόχος που θα μπορούσαμε να θέσουμε ενώπιον μας είναι να δούμε αν υπάρχει μια δυνατότητα. Παρόλα αυτά, τα κράτη-μέλη με όλες τις τεράστιες εντάσεις που υπάρχουν πιέσεις στους δικούς τους προϋπολογισμούς να, να κερδίσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν κάτι παραπάνω στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διότι θα είναι πεισμένα ότι υπάρχει κατάσταση win-win ότι κάτι περισσότερο μπορούμε να, και μπορούν να κερδίσουν από ότι αν μένανε στα εθνικά πλαίσια και αυτά πρέπει πολύ σοβαρά να τα συζητήσουμε όλα και καταλήγω στην τελευταία μου παρατήρηση εδώ έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον πλειοψηφικά από το 2007 προς, ε, εγκρίναμε τις δημοσιονομικές προοπτικές και είπαμε ότι θα υπάρχει ενδιάμεση αναθεώρηση, αναθεώρηση, mid-term review και θα δούμε πώς αυτά όλα δαπανώνται, πώς προχωράμε, όλα αυτά θα σταθμιστούν και θα μετρηθούν υπήρξε επίμαχο θέμα σε σχέση με αυτό. Όμως όλο και λιγότερο συμφέρον και ενδιαφέρον έχει το, το Συμβούλιο. Το μεγάλο ερώτημα είναι θα καταλήξουμε σε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση και πώς. Εκρεμεί το θέμα. Είναι μετέωρο. Και υπάρχει ο κίνδυνος όλο και λιγότερο να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε σε επίκαιρα αιτήματα και απαιτήσει. Αφενός τι θα κάνουμε με τις ρεαλιστικές αυτές εκτιμήσεις, αλλά και με τις πολιτικές αναγκαιότητες να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αν θέλουμε να πάρουμε τους στόχους μας στα σοβαρά, ε, τότε θα χρειαστεί πραγματικά μια ανοιχτή συζήτηση για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, διότι διαφορετικά τους επόμενους μήνες θα τροχοπεριθούν τα πράγματα και αυτό θα είναι ιδιαίτερα δραματικό. Merci, Σε ευχαριστώ. Σαλβαδόρ Γκαρίγα ζήτησε τον λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, γιατί Άλλοι συνάδελφοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για την έκθεση του Ράιμερ Μπέγκε και την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι μέρος της συζήτησης <clears throat> που σε σχέση με το ποια είναι τα όρια και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τι θα γίνει στο μέλλον. Μέρος αυτής της συζήτησης θα έπρεπε να το μεταθέσουμε προς μια νέα δομή εσόδων. Μια νέα δομή εσόδων που δεν θα σήμαινε δημιουργία νέων πόρων, κοινοτικών πόρων, αυτό θα ήταν μια αντίφαση με τις πολιτικές της λιτότητας. Ωστόσο όμως περισσότερο να αντισταθμίσουμε, να εξισορροπήσουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ευρωπαϊκό κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτή η ιδέα που είναι αυτονόητο και εμφαίνεται σε κάποια έγγραφα του ίδιου του Λαμασούρ ή και του ε, συναδέφου, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια συνεισφορά από πλευρά τη Επιτροπή προπολογισμών για τη μελλοντική συζήτηση που θα διεξαχθεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ανάγκη να καταδειχθεί ότι κάποια πράγματα που γίνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να σημαίνουν μια εξοικονόμηση κονδυλίων από ό,τι αν γινόντουσαν από τα κράτη-μέλη. Είναι ο μόνο τρόπο που θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μα στο μέλλον και να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι νέε προκλήσει και ανάγκε για τα νέα προγράμματα πράγματα που όπως πολύ καλά είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι σαφές ότι δεν υπάρχει επαρκές περιθώριο ελιγμών από πλευράς κονδυλίων. Δεν θα ζούμε όλα τα χρόνια από τα πλεονάσματα της Γεωργίας. Το ξέρουμε ήδη ότι το 2011 και στα ε, συνεχόμενα έτη δεν θα μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό το μόνο που πρέπει να αναζητηθεί είναι μια νέα ισορροπία μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και μάλιστα στο εγγύς μέλλον να εξευρεθεί αυτή η ισορροπία. Ε, Quelques commentaires de mon côté. μερικά σχόλια δικά μου τώρα. Φυσικά η σημερινή συζήτηση είναι κάπως εκτός φάσης σε σχέση με την κατάσταση που ζούμε εδώ και 48 ώρες. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για το θέμα αυτό όπως μιλούσαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πώς πρέπει να μιλήσουμε. Παράδειγμα, Σήμερα η εντύπωση που έχουμε είναι θερμό. Μετά την οξία αυτή η κρίση και το πολύ θεματικό πράγμα που φαίνεται ότι καθυσίχασε κάποιες αγορές. Η εντύπωση είναι ότι όλες οι χώρες μας θα είναι υποχρεμένες να έχουμε πολύ αυστηρές πολιτικές προπολογισμού. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να ζητήσουμε όλοι οι προπολογισμοί να μειωθούν εκτός από τον ευρωπαϊκό. Αυτό ως απεισιόδοξο. Και όλοι διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να συνοδευτεί αυτό το πρόγραμμα λιτότητας για ένα-δύο χρόνια να έχουμε έναν προπολογισμό της κοινότητας χωρίς αύξηση. Υπάρχει όμως και διαφορετική και άλλες λύσεις, δυνατότητες. Μέχρι πριν από τρεις μέρες όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και όλοι οι νομικοί μας εξηγούσαν ότι η Ένωση δεν μπορεί να χρεωθεί. Και εγώ ίδιος το έλεγα. Λάθος. Το άρθρο 122 δεν προέβλεπε μη δυνατότητα δανεισμού. Προέβλεπε δυνατότητα να δοθεί οικονομική ενίσχυση της Ένωσης. Οικονομική υποστήριξη της Ένωσης. Ελήφθη η απόφαση και η νομική μας αποδεικνύουν ότι συμφωνεί απόλυτα με τις συνθήκες. Αυτός βέβαια είναι ο ρόλος των νομικών. Οι νομικοί μπορούν να αποδείξουν ότι όλα τα πάντα είναι πάντα δυνατά αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Βέβαια, αυτή είναι η καλή νομική και από την πλευρά υπάρχουν καλοί πολιτικοί που θα του πούνε να έτσι να κάνετε για να παραβιάσουμε τι συνθήκε για να ε, ε, μας εξηγήσουν ότι δεν παραβιάστηκαν οι συνθήκες. Τώρα λοιπόν είναι δυνατό η Ένωση να δανειστεί για να δανείσει έναν κακοδιαχειριζόμενο κρατικό προπολογισμό. Και πολιτικά θα εξηγηθεί ότι αντίθετα η Ένωση δεν μπορούσε να δανειστεί για να δανείσει στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ο οποίος είναι ο πιο καλά διαχειριζόμενος ο κοινωτικό σε σχέση με όλου του άλλου. Γιατί όπω είπε η Άν υπάρχουν ένα σωρό προγράμματα μέσα γεμάτα μέλλον. Τα πιο υγιή προγράμματα για την οικονομική ανάπτυξη. Για να συνοδευτεί έξυπνα ένα πρόγραμμα ανάκαμψη που δεν είναι ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που τιμωρεί, δεν είναι πρόγραμμα λιτότητα, αλλά είναι ένα πρόγραμμα μέλλοντο. Αυτή ήταν η πρόταση της Λευκής Βίβλου Ντελεόρ. Και όλοι είπαμε Ω, δεν γίνεται, ο ευρωπαϊκός προπολογισμός κλπ. Κακός. Από σήμερα ο ευρωπαϊκός προπολογισμός υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί σε έγκλημα 60 δις. Αυτό αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό είπα πολύ προσοχή στα εκτός προπολογισμού, γιατί θα μας πούνε, μα δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ναι, είναι κοινωτικό, αλλά δεν είναι ο προπολογισμό. Πώς δεν είναι ο πού είναι και από τη στιγμή που φυσιολογικά θα πρέπει να πούμε ναι, είναι ο κοινωνικό προβλησμός, να θέσουμε το πολιτικό ερώτημα. Η Ένωση έχει δικαίωμα να δανειστεί μόνο για να δανείσει σε ένα χρόνο μέρο που κακοδιαχειρίζει τον προπολισμό ή για να χρηματοδοτεί ή δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει πολιτικέ που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αλλιώ. Δηλαδή τι τελευταίε μέρε όλα αυτά που έγιναν αλλάζουν τα δεδομένα. Και μπορούμε να έχουμε είτε μια θλιβερή απεσιόδοξη λύση και κατάσταση στην οποία όλοι άβουλα θα συμμετάχουμε και θα ζήσουμε κατάσταση ανορεξίας ή σε κάτι θετικό. Να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Μπορεί η έργα να χαμογελάσει όταν θα το ακούσει, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ να κάνω την έργα να χαμογελάσει. Θα μπορούσαμε να πούμε, αν δεχτούμε την ιδέα να μοιραστούμε τους ρόλους στη χρηματοδότηση των κατά προτεραιότητα πολιτικών μεταξύ των κρατικών προπολογισμών και ημών με ΙΤΑ. Και θέσαμε το ερώτημα στους εκπροσώπους, θα θέσουμε μάλλον το ερώτημα στους εκπροσώπους ε, βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια, στην Επιτροπή Προπολογισμού. Θα τους πούμε. Εμείς υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού θα κάνουμε μια προσπάθεια λιτότητας, δεν θα αυξήσουμε. Εκτός από ένα τομέα. Εμπιστευτείτε μας αυτή την ευθύνη γιατί είναι στις αρμοδιότητες της Λισαβόνας και συμφωνεί με όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες που πήρε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εδώ και τρία χρόνια. Περιβάλλον. Ενέργεια και περιβάλλον. Υπάρχουν προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, επαναπροσανατολισμό της κατανάλωσης ενέργειας προς καθαρές μορφές, προστασία περιβάλλοντος, ερευνητικά προγράμματα κλπ να χρηματοδοτήσουμε αυτά με νέους πόρους που θα έχουμε από το 2013 η πώληση με διαγωνισμό των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που θα επιβληθεί στις βιομηχανίες, στις μεταφορές που δυστυχώς εκπέμπουν τέτοιου είδου αέρια. Δεν είναι η πρώτη πολιτική μου προτεραιότητα, αλλά είναι μια επιλογή. Έχει νόημα να το πούμε. Για να καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι από τη στιγμή που όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση πρέπει να δουλέψουμε από κοινού, να βρούμε κοινή λύση, να μοιραστούμε το έργο. Και το Ευρωκοινοβούλιο και ο προπολογισμό της Ένωσης μπορεί να παίξει κάποιο θετικό ρόλο χωρίς να στοιχήσει στο φορολογούμενο και χωρίς να επιβαρύνει το χρέος. Εφιστώ την προσοχή σας, συνάδελφοι, στο ότι σήμερα είναι δύσκολο να καταλήξουμε κάπου. Είναι δύσκολο να πούμε σήμερα τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίθετα, Έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού που είναι η προφορική ερώτηση. Προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης ολομέλειας του Μαΐου 2. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα τον Ιούνιο να καταλήξουμε κάπου. και αν όλα πάνε καλά, η Κομισιόν μέχρι τότε μας έχει προτείνει, βλέπω ο Γενικός Διευθυντής χαμογελάει, δεν θα τον βασανίσω για να μας απαντήσει, μας πρότεινε άλλα κείμενα. με βάση τις επιθυμίες της Επιτροπής μας. σε θέματα προσαρμογής ή αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν κάποιο θα έγινε να πάρει το λόγο. Ο Ράιμερ βλέπω έγινε να πάρει το λόγο. Πράγματι, οι εξελίξεις που αντιμετωπίζουμε αλλάζουν και κάποιες ε, συζητήσεις εδώ μέσα και τα συμπεράσματα που θα πρέπει να, να βγουν για το τι θα κάνουμε παραπέρα και βεβαίω αυτά τα οποία είχαμε προγραμματίσει πλέον αλλάζουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, οπότε ο Πρόεδρος ε, κάνει πολύ σωστές προτάσεις. Να πω επίσης πως έχει δίκιο ο Γκορνφέρμ πως ε, πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να δούμε πως θα μπορέσουμε πως ε, εφόσον βεβαίως και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις Λισαβόνας δεν αφορούν μόνο την εξωτερική υπηρεσία που είναι και αυτό ένα μέρος του πακέτου αλλά να δούμε τι θα κάνουμε με, επί τη βάση των συζητήσεων με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για το πώς θα προχωρήσουμε με την διατύπωση τροπολογιών ε, επί των προτάσεων της ε, Κομισιόν και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και για το πώς θα αλλάξει η διοργανική ε, συμφωνία. Περιορίζομαι τώρα στην έκθεση για την οποία είμαι υπεύθυνο εγώ για να ξεκαθαρίσω πως όσον αφορά την αλλαγή του πολιετούς πλαισίου χρειάζεται βέβαια σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και να μένουμε σοβαρές συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα γιατί εντάξει ελπίζουμε πως κάποτε θα υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο και μετά θα πρέπει να συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει πως ε, με βάση τη χρονική πίεση θα πρέπει να συμφωνήσουμε και εμείς σε ό,τι πουν χωρίς να το εξετάσουμε. Θα πρέπει να μας πάρουν ε, τελείως ε, σοβαρά στις συζητήσεις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν εδώ πέρα τον Νοέμβριο. Οπότε θα πρέπει να συνοηθούμε εμείς εδώ πέρα για τα ουσιαστικά. Και αυτή είναι η συζήτηση που απαιτείται στα ζητήματα στα οποία θα δώσουμε έμφαση. Ευχαριστώ. Alors, je vous propose maintenant... Σε ευχαριστούμε, Ράιμερ. Ας περάσουμε στα εννέα. Που είναι η κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ έχουμε δύο πτυχές είναι η κινητοποίηση για τεχνική βοήθεια προς την Κομισιόν και το πιο κλασικό ετοιμάτων των κρατών μελών. Μια ανταλλαγή απόψεων, στα γρήγορα. Στην έκθεση της Μπάρμπερα Ματέρε που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εφιστώ την προσοχή των συναδέλφων στο αίτημα της ε, κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αίτημα της Κομισιόν, τελείως διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν, διότι αναφέρεται στο άρθρο 8.1 του κανονισμού, όπου το 0,35% του ετήσιου προπολογισμού του Ταμείου πάει για την τεχνική βοήθεια να ελεγχθεί ο μηχανισμός και η χρήση του ταμείου αυτού. Είναι 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Με τους εξή στόχους. Πρώτο, monitoring. Η Κομισιόν προτείνει παράγγες μελέτες για την εφαρμογή της χρήσης αυτού του ταμείου κόστος 250.000 δεύτερον το site internet 240.000 ευρώ δημιουργία μιας βάσης γνώσεων θα γίνει μια μελέτη όπου θα συλλέγονται διάφορα στοιχεία, περιπτώσεις απολύσεων, εμπειρίες εργαζομένων, κόστος 50.000 ευρώ. Διοικητική τεχνική υποστήριξη, δύο συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονες της Κομισιόν και υπεύθυνου του Ταμείου αυτού από τα 27 κράτη για φέτος 70.000 ευρώ. Μετά έχουμε την ανταλλαγή των best practices, συναντήσεις μεταξύ των κρατών μελών με συμμετοχή προσώπων που θα έχουν μαζί τους και εμπειρογνώμονες για να προετοιμαστούν τα αναγκαία κείμενα προκειμένου να ε, προετοιμαστεί το αίτημα του Ταμείου. 200.000 ευρώ. Τέλος έχουμε την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου. 300.000 Δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτή η πρόταση. Ζητήθηκε υποστήριξη από το, ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περιμένουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης που έχει ομάδα εργασίας στις 19 Μαΐου και η ψηφοφορία θα γίνει την 1η Ιουνίου, μία μέρα πριν ψηφίσουμε εμείς. Ιουνίου. Μακάρι να μην υπάρξουν προβλήματα στην Επιτροπή Απασχόλησης και όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, ήδη έχουν γίνει τρία αιτήματα από δύο κρατημέλη για το Ταμείο αυτό. Πρώτο από την Ιρλανδία για τη βιομηχανία κεραμικιά και κρίσταλα. Κρυστάλλινα. 598 εργαζόμενοι. Το νούμερο, το ποσό είναι 2 εκατομμύρια 570.000. Μετά έχουμε ένα αίτημα από την Ισπανία κεραμικά που έχουν σχέση με την οικοδομή 181 επιχειρήσεις, 1.600 εργαζόμενοι, κονδύλι, 6 εκατομμύρια 6,6 εκατομμύρια ευρώ. 6,6 και το τρίτο για την Ισπανία, βιομηχανία, ε, διάφορα προϊόντα πλεκτικής, υφάσματα κλπ. Πολλές επιχειρήσεις, 500 50 περίπου εργαζόμενοι 1,95 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό θα χρειαζόμαστε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σε ευχαριστούμε, Μπαρβαρά. Στάει κανείς το λόγο. Όχι, σε ευχαριστούμε για τη σαφή παρουσίασή σου. Όπως και η Μπάρμπαρα έχουμε δύο διαφορετικά εργαλεία εδώ, νομικά εννοώ. Το ένα είναι για την κινητοποίηση για τεχνική βοήθεια προς την Κομισιόν με ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 2 ε, Ιουνίου, 1η Ιουνίου στην Επιτροπή Απασχόλησης. Μετά έχουμε τα τρία συγκεκριμένα αιτήματα. Ένα από την Ιρλανδία, ένα από την Βαλένθια της Ισπανίας και ένα από την Καστίγια Λαμάνσα Ισπανία. Η Κομισιόν απασχόλησε θα το μελετήσει το Μάιο και θα έρθει σε εμά 21 με 22 Ιουνίου. Ευχαριστούμε την Μπάρμπαρα. Ξέχασα το 6. Προτείνω να μην ασχοληθώ με το 6. Ψυχολογική σημαντική αυλεψία ήταν αυτή, διότι ε. πρόκειται για το διορθωτικό προπολογισμό 4. 2009. Εδώ λέει 10, αλλά μάλλον το 9 είναι. Ναι, ναι, 2010. Διορθωτικό 2010. Με θέμα είναι τα πλεονάσματα του 2009. Έχουμε πλεονάσμα. Μάλιστα. Μπορεί να περιμένει. Ο ζητητής απουσιάζει. Κρίμα. Λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι τα σύννεφο από το ηφαίστειο καθυστέρησαν τον εισηγητή. Αν όλοι συμφωνούμε, θα περιμένουμε. Εκτός αν ο Σαλβαντόρ θέλει να αντικαταστήσει, αλλά το θέμα είναι τον εισηγητή, αλλά το θέμα είναι τόσο πολύπλοκο που σας προτείνω να μην μελετήσουμε σήμερα το 6. Θα έχουμε άλλη ευκαιρία αργότερα. Να το δούμε με στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού και πολιτικού τοπίου. Ο Γκέραν δεν συμφωνεί. Φέρουμε. Πρόεδρε, εσείς ή κάποιος μπορεί να μα πείτε τι επιλογές έχουμε. Νομικά υπάρχει η πιθανότητα, η δυνατότητα να καθυστερήσουμε, να τροπολογήσουμε, ακόμη και να απορρίψουμε. Νομικά, πού βρισκόμαστε. Πρόεδρος. Επειδή ακριβώ και εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω και ο εισηγητής απουσιάζει, γι' αυτό σας πρότεινα να το αναβάλουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποφασίσουμε σήμερα. Γιατί έχω ακούσει πολλά αντιφατικά. Έχουμε τις συνθήκες. Έχουμε το δημοσιονομικό κανονισμό και έχουμε ένα είδο συμπεριφοράς τι είναι, gentleman's agreement, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, μέχρι τώρα το πολιτικά ορθό ήταν όταν η Κομισιόν διαπιστώνει πλεόνασμα, αμέσως το έδινε στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται όμω διαδικασία, χρειάζεται ψήφος του Κοινοβουλίου. Εγώ δεν είμαι, μεγάλο, δεν είμαι μεγάλος νομικός, είμαι απλός άνθρωπος. Και λέω, σε μια δημοκρατία δεν μπορούμε να πούμε ένα θέμα που υπόκειται στην ψήφα του Κοινοβουλίου, πρώτον. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να πει ναι. Τρίτον, εν η ψήφο του Κοινοβουλίου δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Που είναι καθεστώ τύπου Κεντρική Ασία, αλλά δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν το Κοινοβούλιο ψηφίσει, αν χρειάζεται διαδικαστικά, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να πει όχι. Μπορεί να μην έχει δικαίωμα να, τροποποιη... να τροπολογήσει, μπορεί να πει όχι. Ή τουλάχιστον να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τη μέρα που θα πάρει την απόφαση. αλλιώ πρέπει να αλλάξουμε τι συνθήκε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και σα είπα δεν είμαι μέγας νομικό. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς μας μερικές μέρες ακόμα να τις αξιοποιήσουμε για να είναι σαφής για μας η νομική κατάσταση. Στόσο ο Σαλβατόρη θέλει, βλέπω εκεί, θέλει, ψώνει και καλά να πάρει το λόγο. Μόνο για να σας πω, το είπατε εσείς πολύ ευφυώς ότι αυτή η προθεσμία 42 ημερών για να ληφθεί μια απόφαση έγκαιρα στην επόμενη Επιτροπή Προϋπολογισμών θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε αν σύμφωνα με τις μεταβατικές ρυθμίσεις δεχόμαστε, τροποποιούμε ή απορρίπτουμε αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμό 4. Εν πάση περιπτώσει 42 ημέρες είναι και έγκαιρα θα είμαστε για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών όπου όλοι αναμένουμε ότι τα προβλήματα τα οποία έχει το Συμβούλιο με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς θα έχουν αρθεί ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Σαλβατόρ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Θα ξαναδώσω το λόγο στο Σαλβατόρ, που αντικαθιστά το συνάδελφο εισηγητή Πουλτίτη, για το 10 μιλάω, Αναβάλλεται το 10. Α, αναβάλλεται. Δεν υπάρχει μεταφορά. Ωραία. Το 10 έφυγε. Αναβάλλεται. 11. Ενδεχομένως άλλες μεταφορές πιστώσεων. Ο συγκεκριτής έχει φύγει. Δεν έχουμε τίποτα γι' αυτό. 12. Αποφασίσαμε ότι αναβάλλεται, γιατί η συνάδελφος Ανδρεάσεν λείπει. Προθεσμία δεν έχουμε εδώ. Ευτυχώς η Γιούτα είναι εδώ. Γνωρίζει το θέμα της και θα μας παρουσιάσει την κατάσταση του Οργανισμού για την Λειτουργική Διαχείριση Μεγάλων Συστημάτων Πληροφορικής σε θέματα της ε, πληροφορικής γνώμης στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Γιούτα Χάουγκ. Ευχαριστώ. Το θέμα το ξέρω νομίζω αρκετά ε, έτσι ώστε τουλάχιστον να θέσω το ερώτημα το αν θα πρέπει να αποφασίσουμε και να εγκρίνουμε εμείς με την γνωμοδότησή μας αυτό το οποίο προτείνεται η Κομισιόν ε, τον Ιούνιο πέρσι έκανε αυτή την πρόταση να γίνει δηλαδή μία υπηρεσία, ένας οργανισμός ε, που θα κάνει τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων συστημάτων πληροφορικής. Και όπως είπε ο πρόεδρος, μάλιστα στον τομέα ελευθερίας ασφάλεια και δικαιοσύνης, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει το σήμα πληροφοριών Σίγγεν 2, το SIS2 όπως λέγεται, το σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων, το VIS δηλαδή, και το Eurodac. Το σύστημα δηλαδή πληροφορικής για την υποστήριξη και χρήση της συνθήκης ε, του Δουβλίνου. Για άσυλο δηλαδή, αιτήσεις ασύλου από, τρι, από χωρών. Όλα αυτά να πάνε μαζί σε μία υπηρεσία που θα τα διαχειρίζεται. Η υπηρεσία αυτή προτείνει η Κομισιόν θα πρέπει μέχρι το τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών για τις οποίες μόλις μιλήσαμε την Μακρόν να κοστίσει 113 εκατομμύρια ευρώ. Τα λεφτά αυτά μας λέει η Κομισιόν δεν αποτελούν πρόβλημα γιατί δεν επηρεάζεται, δεν επιβαρύνεται πάρα πολύ το υπάρχον περιθώριο γιατί θα πάει από τις τρεις ανάλογες αντίστοιχες γραμμές του προπολογισμού. Κοιτάζοντα λοιπόν εδώ πέρα τα πράγματα, επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να μου απαντήσει η Κομισιόν. Εάν κοιτάξουμε τι είναι στο Eurodac το SIS και το VIS και τα προσθέσουμε, καταλήγουμε στα 401 εκατομμύρια ευρώ. Η δε μελλοντική υπηρεσία θα απορροφήσει τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Τι θα συμβεί με τα υπόλοιπα 288 εκατομμύρια. Τι θα τα κάνουμε. Γιατί προβλέπονται. Πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Και εδώ πέρα παρακαλώ την Κομισιόν για το όνομα του Θεού να μας στηρίξει. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ πως εάν είναι να μιλήσουμε για το μέλλον αυτού του προπολογισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το, την συνέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε το τι σημαίνει αυτό για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Εξήγησα ήδη το τι θα κάνει αυτή η υπηρεσία. Αυτό όμως σημαίνει πώς θα πρέπει να γίνει και πάρα πολύ, θα φύγει μάλλον πάρα πολύ δουλειά από τους εθνικούς προπολογισμούς. Θα ελαφρυνθούν δηλαδή οι εθνικοί προπολογισμοί. Θέλω αυτό το πράγμα να μου το ε, γράψει κάπου η Κομισιόν. Να γνωρίζουμε δηλαδή, αν λάβουμε αυτή την απόφαση, τι εξοικονόμηση υπάρχει στον, στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και να μην λέμε, όπως συνήθως, πώς θα πάει η δουλειά στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όλοι οι υπόλοιποι να λένε «Α, ωραία, συνεχίζουμε εμείς σαν να μην συμβαίνει τίποτα». Το δεύτερο ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Θέλω μια αξιολόγηση αντικτύπου. Τρίτον, η υπηρεσία όταν ξεκινήσει την δουλειά της θα έχει γύρω στα 120 άτομα. 120 άτομα μόνο για αυτή την υπηρεσία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το αντικείμενο εργασίας της, Κομισιόν γίνεται, της ε, υπηρεσίας γίνεται από την Κομισιόν. Τη δουλειά αυτή την κάνει τώρα η Κομισιόν. Αλλά πουθενά δεν βλέπω να υπάρχουν μεταθέσεις. Οι άνθρωποι δηλαδή που κάνουν τώρα αυτή τη δουλειά στην Κομισιόν να πάνε σε αυτή την υπηρεσία. Κάθε άλλο. Ε, λένε πως ε, τέσσερα άτομα της Eurodac και ένας εξωτερικός συνεργάτης θα πάνε σε άλλες υπηρεσίες κομισιών. Ε, όχι, κατά την άποψή μου αυτοί ανήκουν στην υπηρεσία αυτή. Πρώτον. Δεύτερον, αλλά 20 υπάλληλοι και 25 εξωτερικοί συνεργάτες του ΣΥΣ2 και του ΒΙΣ θα πρέπει και αυτοί να πάνε αλλού Κανένας δεν ε, μιλάει για μετάθεση στην υπηρεσία αυτή. Τέταρτον, ε, θα ήθελα να μάθω βεβαίω τι, τι σκέφτεται εδώ πέρα η Κομισιόν. Ξέρουμε τι σκέφτεται, αλλά θέλω να μας το πει η ίδια. Τέλος, αξιολόγηση αντικτύπου, όπου έχει, έχει δεσμευτεί να το κάνει η Κομισιόν και πάντα δηλαδή όταν λέμε ότι θέλουμε μια καινούργια υπηρεσία, να δούμε ποια είναι η προσθέμενη αξία και ποια είναι σε σχέση με την ε, υπάρχουσα υπηρεσία της Κομισιόν. Ε, είναι λίγο παλαιού τύπου αυτή η ε, αξιολόγηση αντικτύπου και είναι λίγο παλαιωμένη κιόλας, είναι τριών ετών. Και εν τω μεταξύ, σε διάφορα μέρη, όχι μόνο στην Επιτροπή Ελευθεριών, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια, πάντα ασκείται κριτική πως έτσι όπως έχει συλληφθεί αν θέλετε και επινοηθεί αυτή η υπηρεσία δεν υπάρχει καμία εγγύηση προστασίας προσωπικών ε, δεδομένων και έχουμε την συζήτηση που ξέρετε για τη μεταφορά δεδομένων και προστασία δεδομένων κτλ. Την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση με τις ΕΠΑ και τουλάχιστον εδώ πέρα εμείς θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον τόσο ευαίσθητοι όσο απαιτούμε από τα άλλα κράτη με τα οποία έχουμε συμβάσεις. Και ταυτόχρονα ήδη τώρα εντάξει η ιδέα είναι παλιά αλλά εντωμεταξύ έχουμε μια ε, υπηρεσία ένα γραφείο πως λέγεται για την στήριξη όσων ζητούν άσυλο. υπάρχει εδώ πέρα κάποια αλληλεπικάλυψη με την υποσύσταση αυτή η υπηρεσία. Πριν κάνουμε λοιπόν την γνωμοδότησή μας για την Επιτροπή Ελευθεριών, χρειαζόμαστε πολλές πληροφορίες από την Κομισιόν και πιθανώς, δεν ξέρω κάποιος συνάδελφος, ε, να έχει και άλλες ερωτήσεις ε, για την Κομισιόν, ε, τις οποίες θα θέλαμε να απαντηθούν. Οι θα θέλαμε να απαντηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Κομισιόν ε, μπορεί να απαντήσει. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το λόγο στο συνάδελφο της Γενικής Διεύθυνσης για την θέματα ελευθερίας, ασφάλειας κλπ. Για να απαντήσει πιο συγκεκριμένα ένα σημείο που ανάφερε η κυρία Χάουγκ εξοικονόμηση ενέργεια όσον αφορά του ανθρώπινου πόρου στην Κομισιόν για δραστηριότητε που θα μεταφερθούν στον οργανισμό. Αυτή την εξοικονόμηση τη χρησιμοποιούμε σε, άλλους, σε άλλα πεδία όπου οι πολιτικέ προτεραιότητες απαιτούν μεγαλύτερη δραστηριότητα. Περισσότερη δουλειά για την Κομισιόν. Και έτσι η Κομισιόν μένει μέσα στις δεσμεύσεις που έχει να μην ζητήσει επιπλέον προσωπικό. Για τα υπόλοιπα επιτρέψτε ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια να μας απαντήσει. Ο κ. Διευθυντής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά ένα προς ένα. Πρώτα απ' όλα για το κόστος. Υπήρχαν δύο ερωτήσεις για το κόστος. Η πρώτη αφορούσε το υψηλό κόστος ε, σε σχέση με τα συστήματα αυτή τη στιγμή και την νέα υπηρεσία και το τι θα γίνει με την εξοικονόμηση σε εθνικό επίπεδο το κόστος ε, αφορά μόνο την σύσταση και τη λειτουργία της ε, υπηρεσίας, αλλά καλύπτει και την λειτουργία των συστημάτων ε, που θα διαχειρίζεται η υπηρεσία, αλλά όχι την ανάπτυξη των συστημάτων που σχετίζονται με τα μέσα και την νομική βάση του κάθε ε, συστήματος ξεχωριστά. Υπάρχει δηλαδή κόστος για την ανάπτυξη του Eurodax και VIS, αλλά είναι σε διαφορετική νομική βάση και νομικό μέσο το καθένα για τους ίδιους λόγους Ε, επειδή θα υπάρξει κάποια διευκόλυνση στα κράτη-μέλη, η απάντηση είναι όχι, γιατί το κόστος ανάπτυξης πάλι καλύπτεται από την νομική βάση των συστημάτων των ίδιων για το Eurodac SIS2 και το VIS, που θα είναι διαφορετική όταν θα είναι επιχειρησιακά τα συστήματα και θα αρχίσει να διαχειρίζεται αυτή η υπηρεσία, γιατί όλο το κόστος τότε θα πάει στην υπηρεσία. Για το δε προσωπικό νομίζω απαντήθηκε ήδη η ερώτηση. Μάλιστα η πρόβλεψη είναι πως όταν θα αναλάβει η υπηρεσία και θα είναι επιχειρησιακή, το προσωπικό της Κομισιόν που τώρα ε, απασχολείται σε αυτό το αντικείμενο θα μειωθεί σταδιακά. Αξιολόγηση αντικτύπου, ναι, έγινε μία αξιολόγηση αντικτύπου, ήταν η βάση της πρότασης αυτής που έχουμε τώρα μπροστά μας. λύση η οποία προτάθηκε και όσον αφορά την ε, νομική βάση και την δομή, αν θα είναι κεντρική ή αποκεντρωμένη, ήταν επίσης αντικείμενο της αξιολόγησης ε, αντικτύπου και η λύση ήταν αυτή ε, που ακολουθήσαμε. Τώρα γιατί να μην το κάνει η Κομισιόν και να το κάνει η υπηρεσία. Ήταν ένα ερώτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ και Υπήρχε μάλιστα μία κοινή δήλωση Συμβουλίου Κοινοβουλίου Κομισιών για την νομική βάση του ΣΥΣ και του ΒΙΣ που ζητούσε την υπηρεσία συγκεκριμένα γιατί το Κοινοβούλιο τότε, το Συμβούλιο και η Κομισιόν αλλά και η μελέτη που διαπίστωσαν πως μόνο μία υπηρεσία μπορούσε να το διαχειριστεί και όχι τα κράτη-μέλη, ούτε οι Κομισιόν ε, θα μπορούσαν ε, να λειτουργήσουν τέτοια συστήματα πληροφορικής που είναι κρίσιμα για την ε, αποστολή που χρειάζεται Τώρα, για την προστασία των δομένων το συζητήσαμε εντατικά με την Επιτροπή Ελευθεριών η απάντηση είναι πως οι κανόνες είναι σαφείς ε, στον κανονισμό και στα τρία νομικά βάσα και η ίδια υπηρεσία βεβαίως ε, θα τηρήσει πλήρως τον ε, σχετικό κανονισμό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασία Δεδομένων θα έχει πλήρη εξουσία επί της νέα αυτής υπηρεσία. Επίσης δεν θα είναι χρήστη των δεδομένων με καμία μορφή είναι αυτή η υπηρεσία. Θα διαχειρίζεται μόνο τα συστήματα. Τα κράτη-μέλη θα είναι οι ιδιοκτήτε των δεδομένων. Απλά το σύστημα θα διαχειρίζεται το, το υλικό που διασφαλίζει το ότι θα μεταδίδονται τα δεδομένα. Επίσης υπήρχε μια ερώτηση για την διαλειτουργικότητα. Αυτό ήταν κάτι που το συζητήσαμε στην Επιτροπή ε, Ελευθεριών ως κάτι το σημαντικό. Επ' αυτού θα έλεγα πως δεν προβλέπεται, για την ακρίβεια μάλιστα ρητός απαγορεύεται από την νομική βάση και θεωρούμε πως είναι μια σημαντική διασφάλιση για να προστατευθούν ε, τα προσωπικά δεδομένα στο σύστημα τώρα αλληλεπικάλυψη με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σύλλο. Όχι, δεν υπάρχει καμία αλληλεπικάλυψη, δεν υπάρχει τίποτα στην εντολή, στις αρμοδιότητες ε, της υπηρεσίας ε, αυτού, του, αυτής της υπηρεσίας και της υπηρεσίας για το άσυλο. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ κυρία Συγγήτρια. Λοιπόν, πρέπει πραγματικά για να αποσαφινιστούν τα πράγματα να ξαναρωτήσω επερώτηση. Είναι απόλυτα σαφές, εντάξει, πρέπει εδώ να πω, είναι και άλλη μία φορά ένα παράδειγμα για τα όσα ψευδώς ε, ισχυρίζονται από την Επιτροπή. Είχαν πει από πλευρά της επιτροπή ο κύριος Λεβαντός ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στελεχών. Είναι απλό λοιπόν να επιτευχθεί αυτό. Αν ε, κάνουμε outsourcing σε πάσης φύσεως ε, διοικητικό έργο και υπάρξει μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ε, του προσωπικού, ε, τότε φυσικά όλο μεγαλύτερο θα γίνεται το στελεχειακό δυναμικό των ε, υπηρεσιών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει πλέον, λέει, άλλα στελέχη. Αυτό είναι ένα ψεύδος, αλλά δεν ευθύνεστε εσείς γι' αυτό. Είσαστε εκείνος ο οποίος θα ακούσει αυτές τις επικρίσεις. Ε, όμως ρώτησα πολύ συγκεκριμένα για τις εξοικονομήσεις που θα υπάρξουν από πλευρά των κρατών μελών όταν θα λειτουργεί η υπηρεσία. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με τα κονδύλια τα οποία πρέπει να κινητοποιηθούν για να υπάρξει η πρικοδότηση για την υπηρεσία, για να υπάρξει η ανάπτυξη των συστημάτων Τεχνολογία ε, τεχνολογίας ε, και πληροφορικής. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς, ε, είπατε μόλις πριν ότι τα κράτη-μέλη λέει δεν θα έχουν εξοικονόμηση κονδυλίων. Ε, τότε λοιπόν Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, να υπάρξει η ίδρυση και λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, αν δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά πρόσθετη δαπάνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορούμε να το δικαιολογήσουμε κάτι τέτοιο εφόσον όλα λειτουργούν όπως ε, και πριν και όπως ε, τα ξέραμε και μάθαμε ότι με το κέντρο στη Γαλλία <clears throat> εκεί όπου θα συλλέγονται τα στοιχεία και μετά θα υπάρχει ε, το backup σε άλλη έδρα. λοιπόν, πρέπει αυτό να το δούμε. Το ερώτημά μου είναι, αληθεύουν πραγματικά όλα αυτά τα οποία εσείς είπατε, δεν θα υπάρξει καμία εξοικονόμηση κονδυλίων για τα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει τώρα να το απαντήσετε κύριε. Αν πείτε ότι δεν μπορώ να απαντήσω, πρέπει πρώτα να πληροφορηθώ και να κάνουμε μια αξιολόγηση πρώτα για να αποσαφινιστεί, εντάξει το δέχομαι. Αλλά αν μου λέτε τώρα, εδώ και τώρα, ότι α, εντάξει, αυτή η υπηρεσία μόνο κάποιο διοικητικό έργο θα έχει και δεσμεύεται αποκλειστικά σε σχέση με τις εντολές που τις δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίποτα άλλο. Έτσι όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νομικές βάσεις με τα τρία συστήματα τα οποία θα λειτουργήσουν, ε τότε είμαι κατά μια υπηρεσία. Θα είναι μια εκτελεστική υπηρεσία αν ισχύουν αυτά τα οποία εσείς ισχυρίζεστε. Διαρωτώ με, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε λοιπόν μια εκτελεστική υπηρεσία για αυτά τα τρία συστήματα. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν έγινε αυτό. Έχουμε εντωμεταξύ αυτά τα δύο μέσα, αυτά τα δύο εργαλεία. Γιατί τώρα λοιπόν, αν δεν μπορούν τίποτα άλλο να κάνουν παραδικητικό έργο, <clears throat> μια και πρόκειται για εκτελεστική μορφής ε, ε, δραστηριότητα, γιατί λοιπόν εδώ δεν ε, ελήφθη η πρόνοια μια εκτελεστική επιτροπή. Ευχαριστώ. Très Νομίζω, ότι η πολιτικό και οικονομικό, δημοσιονομικό πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η πρόταση. Σα ε, επιθυμίζω και εμεί τη μα γεγονομοδότηση. Η αρμόδια επιτροπή είναι η ΓΙΜΠΕ e, Ελευθεριών. Είναι νωρί να μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα. Πρόθεση της εισηγήτριας είναι να μας προτείνει ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης αρχές Ιουνίου να το συζητήσουμε. Και μετά βλέπουμε ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα της ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστούμε τη Ιούτα και μας μένει το 14 μόνο. Σύστημα έγκυρες προειδοποίησης για τα γεωργικά. Ξέρετε ότι η Κομισιόν, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, περιοδικά μας ε, παρουσιάζει την κατάσταση καταναλώσεως των πιστώσεων, ταμείο εγγυήσεων, ΦΕΟΓΚΑ. Πήραμε την πρώτη έκθεση για το 2010, πρώτο τρίμηνο. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σημαντικός είναι ο προπολογισμός για τη γεωργία και τη μερίδιο έχει στον κοινωτικό προπολογισμό. Με πολύ προσοχή λοιπόν θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Λαβία, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία μικρή διόρθωση σε αυτό που είπατε. Γιατί αυτό το early warning και τα στοιχεία που πήραμε αφορούν μόνο τον πρώτο μήνα του 2010, δηλαδή μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Οι επιστροφές προ τα κράτη-μέλη ξεπέρασαν τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν για τον προπολογισμό 2010 κατά τα 33,8 εκατομμύρια. Έσοδα με ειδικό προορισμό 483,8 εκατομμύρια από διορθώσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα λόγω παρατυπιών, υπέρβαση στην ποσόστοση γάλακτος κλπ. Προβλέπονται όμως άλλα 305 εκατομμύρια ευρώ με συγκεκριμένο προορισμό έσοδα. Αυτό που με παραξενεύει και ρωτώ την Κομισιόν αφορά την παρέμβαση στην αγορά. Η χρήση των πιστώσεων για παρεμβάσεις στην αγορά ήταν μικρότερο κατά 70 περίπου εκατομμύρια ευρώ από ό,τι είχε προβλεφθεί. Όπως προβλέπει το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, αυτή η διαφορά για την Κομισιόν που οφείλεται. Και πώς γίνεται σε μια περίοδο που σε όλη την Ευρώπη είδαμε ένα σωρό διαμαρτυρίες αγροτών λόγω των τιμών των προϊόντων που είναι πολύ πιο κάτω από το κόστος παραγωγής, σιτήρα, γάλα, μεσογειακά προϊόντα, όπως το σκληρό στάρι, το λάδι, να έχουμε ένα υπόλοιπο που δεν χρησιμοποιήθηκε για την παρέμβαση στην αγορά. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε τιμές πολύ πιο κάτω από το κόστος παραγωγής και από την άλλη έχουμε ποσά κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ερώτημα προς την Κομισιόν. Άμεσες ενισχύσεις. Ποσοστό χρήσης των πιστώσεων. Μείωση γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ και θα ήθελα να το επιβεβαιώσει η Κομισιόν. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έγιναν οι πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων, οι ενιαίες πληρωμές προς την Ελλάδα, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που έπληξε τη χώρα και που φυσικά σήμανε και μπλοκάρισμα και των γεωργικών δαπανών, άρα και μεταφορές χρημάτων υπέρ των γεωργών. Δηλαδή, θα ήθελε η Κομισιόν να μα πει. Να μας πει κάτι παραπάνω. Πρώτον, για τις παρεμβάσεις στην αγορά και γιατί σε μια περίοδο που οι τιμές είναι τόσο χαμηλές έχουμε κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν και απ' την άλλη αν επιβεβαιώνει το ότι τα κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις άμεσες πληρωμές οφείλονται στο ότι δεν δόθηκαν τα ποσά στους Έλληνες γεωργούς οι οποίοι ζουν και οικονομική και κοινωνική δυσκολία και επιπλέον έχουν και μπλοκάρισμα των πληρωμών, των, των άμεσων πληρωμών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, για να δούμε ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις εύστοχες ερωτήσεις του εισηγητή μας. Ποιος από την Κομισιόν. Γεωργία. Τμήμα Γεωργίας. Ο κύριος Γεωργία θα μας απαντήσει. Σύντομα, Πρόεδρε. Μπορείτε να πείτε το όνομά σας, παρακαλώ, να μας πείτε. Είμαι ο Σμόκη και εργάζομαι στην ε, Γενική Διεύθυνση Επιτροπή. Όσον αφορά το θέμα της Ελλάδας, στην Ελλάδα είχαμε ένα πρόβλημα με τα συστήματα πληροφορικής πέρυσι, όπου πραγματικά οι γεωργοί δεν μπορούσαν να περάσουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά όπως προβλεπόταν. Και για ελεγκτικούς σκοπούς δεν θέλαμε να επιτρέπονται οι πληρωμές προς την Ελλάδα μέχρι ότου να μπορούμε να ελέγξουμε τις αιτήσεις τους. Γι' αυτό υπήρξε καθυστέρηση. Και τώρα έχει υπάρξει η πληρωμή μετά τον έλεγχο σύμφωνα με τον ε, κανονισμό και τις διατάξεις. Υπήρξε μια καθυστέρηση σε σχέση με την κατάσταση που οφειλόταν στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις δαπάνες για την αγορά, αληθεύει, υπάρχει μια μικρή ε, υποχρησιμοποίηση σε σχέση με τα 75 εκατομμύρια που οφείλεται σε δύο λόγους. Στο ε, εγχείρημα αυτό, η, ας το πω έτσι, ταχύτητα ήταν, πιο, ε, ήταν βραδύτερη, οι ρυθμοί ήταν βραδύτεροι από ό,τι είχαν προβλεφθεί. Τώρα όμως ωστόσο 96% έχουν ε, λειτουργήσει σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Υπήρξε μια προσωρινή καθυστέρηση, ναι, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατόν για τα κράτη-μέλη να το ε, επανεξετάσουν. Για τον τομέα το γαλακτοκομικό δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι αυξήθηκαν οι τιμές του γάλακτος και των γαλακτοκομικών για το οποίο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσε ε, την δυνατότητα της παρέμβασης ε, και της επιστροφές από τις εξαγωγές. Αυτή είναι η λόγη. Ευχαριστώ. Monsieur rapporteur, pas d'autres remarques. Δεν έχει καμία παρατήρηση ο εισηγητή. Ωραία, σε ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε την ημέρησα διάταξη. Σα θυμίζω ότι η επόμενη συνάντησή μα είναι την 1η και 2 Ιουνίου. 1η Ιουνίου, πολλή δουλειά. Το πρωί έχω μια ακρόαση από κοινού με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Το απόγευμα, κοινή συνεδρίαση εργασίας με τις ε, επιτροπές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και 2 Ιουνίου τακτική συνεδρίαση. Κλείνει η συνεδρίαση, ας μείνουν οι συντονιστές για να αρχίσει αμέσως η συνεδρίασή μας για να χρησιμοποιήσουμε και τους διερμηνείς.